Καλησπέρα σας. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λοιπόν τις εργασίες μας. Και λόγω του ότι όπως γνωρίζετε έχουμε μόνο δύο ώρες ε, στην ε, διάθεσή μας, ε, γιατί μετά θα έχουμε μια κοινή συνεδρίαση της ΙΤΡΕ και της Επιτροπής Μεταφορών και επομένως μάλιστα θα πρέπει να φύγουμε και από αυτή την αίθουσα και να πάμε σε μια άλλη. Έχουμε ε, τρεις διαφορετικές στιγμές ε, στην ε, συζήτησή μας. Θα έχουμε την κυρία Τζαβέλα η οποία είναι η συγγήτρια ε, για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα το οποίο αφορά την, τις διεργασίες που αφορούν την ενέργεια μέχρι το 2050 και τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες αυτές μέχρι το 2050. Τρεις διαφορετικές φάσεις λοιπόν συζήτησης στη διάρκεια των οποίων θα μιλήσουμε για την τεχνολογική έρευνα και για την ανάπτυξη για την οικονομία, αλλά επίσης και για την καινοτομία. Ε, είναι λοιπόν θέματα τα οποία συνδέονται απολύτως μεταξύ τους και έχουν και τα τρία μεγάλη σημασία. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο σκέλος σε αυτό το πρώτο σκέλος θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς θα διαγραφεί το σενάριο μέχρι το 2050 ε, και θα δώσω αμέσως το λόγο στην συνάδελφο Νίκη Τζαβέλα, η οποία είναι η συγγήτρια για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα κάνει λοιπόν την εισαγωγή κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους ομιλητές που έχουμε σε αυτήν την σημαντική ακρόαση και δεύτερον όλους εσάς οι οποίοι ήρθατε για να ακούσετε την ακρόαση αυτή. Οι δικές μου οι απόψεις σας έχουν επικοινωνηθεί ε, μέσω του ε, σχεδίου της αναφοράς που σας έχω στείλει. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα ήθελα να πάρω περισσότερο χρόνο και θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να δώσω το λόγο στους συναδέλφους μου οι οποίοι έχουν γνωμοδότηση από τις άλλες επιτροπές. Στο τέλος της ακρόασης θα πω δύο λόγια. Σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στους συναδέλφους μου που έχουν τη γνώμη από τις ε, άλλες επιτροπές, γνωμοδότηση από τις άλλες επιτροπές. Ευχαριστώ. Allora, allora, la prima, il primo intervento... Πρώτη παρέμβαση, Σάρου Βόλσκι, από την ΑΦΕΤ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά την εξέταση του οδικού χάρτη για την ενέργεια μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η ενέργεια δεν είναι ένα απλό προϊόν της αγοράς, γιατί είναι και μια πραγματικά εξωτερική πολιτική. Και έτσι την χρησιμοποιούν και οι εταίροι μας. Οπότε το θέμα της ασφάλειας ενεφοδιασμού ε, είναι εύλογες και φυσικά θα μας ενδιαφέρουν και νέες καθαρότερες μορφές ενέργειας, αλλά οι προοπτικές μας για την ενεργειακή μας πολιτική μέχρι το 2050 δεν θα πρέπει να ε, απομακρύνεται από τις εξωτερικές πτυχές της ενεργειακής πολιτικής. Δεν έχουμε μόνο τις αντιδράσεις της Gazprom στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ομότυπο των δραστηριοτήτων της Gazprom στην ε, επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ε, ουσιαστικά ε, η παρέμβαση του Πούτιν ε, ε, εμπόδισε τις ρωσικές επιχειρήσει να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι που δείχνει ότι η Γκασπρόμ είναι όργανο εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Πέραν τη ειδική αυτή περίπτωση όμω, θα πρέπει να δούμε και άλλου πιο αποτελεσματικού τρόπου για να εμπλέξουμε στρατηγικά του εταίρου μα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Να διευρύνουμε τι ε, νομοθετικέ μα διατάξει να προωθούμε το κράτο δικαίου και να δημιουργούμε συνθήκε ε, ίσου ανταγωνισμού, ισότιμου ανταγωνισμού με του ε, γειτονέ μα. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με την αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων που ήδη διαθέτουμε στην εξωτερική μα πολιτική. Για παράδειγμα, την, το χάρτη, τη χάρτα για την ενέργεια, τη συνθήκη για την ενέργεια ή επεκτείνοντα και εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης του μηχανισμούς για τον άνθρακα. Επίσης, τα θέματα ε, προμήθειας και διέλευση ενέργειας προϋποθέτουν ε, προβλεψιμότητα, σταθερότητα και μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επίσης, οι προβλέψεις αυτές δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων που έχουν στρατηγική σημασία όπως είναι το Ναμπούκο. Η πολύ σημαντική είναι και η περιφερειακή συνεργασία για να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά μας και την ανταγωνιστικότητά μας ακόμη και σε περίπτωση που δεν ε, υλοποιηθούν οι στόχοι μας για το κλίμα, κάτι που δεν λαμβάνεται υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε αυτό το roadmap ε, όχι σε 100% ασφαλή πορίσματα, για να το πούμε κατά φημισμό. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν και ένα εναλλακτικό σενάριο, σε περίπτωση που το αρχικό σενάριο δεν υλοποιηθεί μέσω πρόθεσμα. Και για παράδειγμα θα έχουμε μεταβατικά καύσιμα, όπως είναι το σχιστολιθικό αέριο. Για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα των πολιτικών ενέργειας και κλιματικών αλλαγών της Ένωσης, καθώς και για τη συνοχή και την αξιοπιστία της εξωτερικής μας πολιτικής, χρειαζόμαστε μια σφαιρική προσέγγιση. Θα πρέπει να ευθυγραμμίζουμε την ενεργειακή μας πολιτική και με άλλες διαστάσεις των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης, όπως ασφάλεια, γυτνίασης, ανάπτυξης, εμπορίου. Χρειαζόμαστε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των θεσμικών οργάνων, ε, Συμβουλίου Επιτροπής και ΕΕΔ. Και αυτά είναι τα βασικά σημεία που περιλαμβάνει η γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ για τον ε, οδικό χάρτη του 2050. Στόχος μας είναι να εντάξουμε την ενέργεια στους ε, κανόνες της αγοράς. Φυσικά με στόχο μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, α μην ξεχνούμε ότι η ενέργεια αποτελεί ένα στο τμήμα τη εξωτερική μα πολιτική ήδη από σήμερα. Ευχαριστώ. Εκ μέρου τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, η κυρία Γιόρταν. In, uh, Ευχαριστώ. Καταρχήν να καλωσορίσω τους ε, Σλοβαίνους δημοσιογράφους που παρακολουθεί τη δημόσια κρόαση. Έτσι ελπίζω ότι και οι συμπολίτε μας θα ενημερωθούν για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί η αγορά της ενέργειας δεν είναι κάτι εικονικό, κάτι ψηφιακό, αφηρημένο και αόριστο, είναι κάτι που επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Στη γνωμοδότηση που κατήρτησα, περιορίστηκα φυσικά στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τις κλιματικές αλλαγές, την ποιότητα του αέρα, την εμπορία εκπομπών και την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος ήταν ανέκαθεν κινητήριο μοχλός της περιβαλλοντικής πολιτικής, όχι μόνο εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επίγνωση βέβαια της ε, κρίσης που διανύουμε και των προβλημάτων που υπάρχουν στις επενδύσεις, στις απώλειες ανταγωνιστικότητας, απώλειες θέσεων απασχόλησης. Πάντως συμφωνούμε ότι βιώσιμη ανάπτυξη είναι η απάντηση και στην κρίση. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ, όπως ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών, αναζήτηση νέων πηγών ενέργειας, ε, αποδέσμευση, απομάκρυση από τον άνθρακα και εναρμόνιση της περιβαλλοντικής μας πολιτικής με την περιβαλλοντική πολιτική των υπόλοιπων χωρών του κόσμου που είναι πολύ λιγότερο φιλόδοξη. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει να υλοποιήσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει όμως ε, κάτι τέτοιο να γίνει με ταχύς ρυθμούς. Θα πρέπει να επισπεύσουμε τις διαδικασίες ε, που είχαμε αποφασίσει στο παρελθόν, το 2008. Επίσης, η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση ε, των πολιτικών μας για την τεχνολογία και τις υπηρεσίες. Γι' αυτό και στην γνωμοδότηση θέτουμε ένα πολύ σαφή στόχο. Δηλαδή, τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και σημαντικά ορόσημα που θα πρέπει να υλοποιούμε μέχρι το 2050 εκ μέρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, κυρία Κολάρσκα Βομπίνσκα. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, που η Κομισιόν έχει προτείνει μελλοντικά ε, σενάρια και είναι καλό να μην έχουν έτσι, χαρακτήρα δετερμινιστικό, ε, να είναι ανοιχτά στην συζήτηση και ελπίζουμε ότι η δική μας συζήτηση, τα δικά μας σχόλια και οι δικές μας συστάσεις θα συμπεριληφθούν εν τέλει. Για να ξεκινήσει όμως τέτοια συζήτηση στις περιφέρειες και ε, για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε τους πολίτες θα πρέπει να έχουμε μια ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο ε, θα ε, επηρεάσουν τα σενάρια αυτά τους πολίτες. Κάθε χώρα μέλος είναι διαφορετική και θα πρέπει να ακολουθήσει το δικό της δρόμο προς το 2050. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό ο οδικός χάρτης να έχει έχει προσέγγιση βάσει μεμονωμένων χωρών μελών. Αυτό το γεγονός κατέστη σαφές στην ε, πρώτη ε, αναθεώρηση του οδικού χάρτη, αλλά δεν περιλαμβάνεται στην ίδια την έκθεση. Δεύτερο σημείο, το οποίο είναι σημαντικό για την Επιτροπή ε, περιφερειακών ε, ζητημάτων ε, είναι το εξής, ε, ότι θα πρέπει όλες αυτές οι αποφάσεις να στηριχτούν από αποφάσεις περί του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να υπάρχουν για όλα τα σενάρια της ενέργειας που να μπορούν να στηρίξουν, εν πάση περιπτώσει, οικονομικά τα προγράμματα αυτά, αλλά με την προϋπόθεση ότι τα προγράμματα αυτά προωθούν ακολουθούν τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Δηλαδή, να μην χρησιμοποιήσουμε ε, να, να, να χρησιμοποιήσουμε χρήματα παίρνοντας από τη μία τσέπη για να γεμίσουμε την άλλη τα σενάρια για, την, για τον οδικό χάρτη του 2050 δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν εάν δεν υπάρξουν ε, οι απαραίτητες ε, ε, ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει αποκεντρωμένη πράσινη οικονομία εάν σε περιφερειακό επίπεδο δεν έχουμε τα FEE e, grids κτλ. Ε, τέλος, ε, θα ήθελα να καλέσω, ε, να κάνω έκκληση μάλλον, έτσι ώστε το βάρος που θα κληθούν να σηκώσουν οι διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι ισόρροπο έτσι ώστε από τη μία πλευρά οι περιφέρειες να διασφαλιστούν όσον αφορά την ενέργεια, από την άλλη πλευρά να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Σμιτ από την ΙΜΚΟ είναι ο τελευταίος παρεμβαίνων. Είναι εδώ ο συνάδελφος Σμιτ. Όχι δυστυχώς. Ε, επομένως μπορούμε να περάσουμε αμέσως στο πρώτο τμήμα των ε, παρά εισηγήσεών μας. Τον λόγο έχει ο κύριος Γκέρτ Φωστιέ από τη ZDF για 10 λεπτά. Thank you, Well, first of all, I would... Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαρτόρη. Θα ήθελα ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις θέσεις μας για την αποδέσμευση της ευρωπαϊκής οικονομίας από τον άνθρακα. Θα ήθελα να εστιαστώ στην παρουσίασή μου σε κάποιες ε, διαφάνειες και κυρίως να αναφερθώ στα κύρια προβλήματα, στα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, στις δυσκολίες που παρατηρούμε κατά την ανάπτυξη των εξωτερικών σενάριων που κυκλοφορούν ως προς την αποδεσμεύση από τον άνθρακα και μια μελέτη που έχουμε κάνει εμείς στην εταιρεία μας. Θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέπετε να σας ε, παρουσιάσω, να σας καθοδηγήσω στις ε, θέσεις που έχουμε περιλάβει σε κάποιες διαφάνειες για το θέμα αυτό της αποδέσμευσης από τον άνθρακα. Καταρχάς κάποια εξωτερικά σενάρια που θα ήθελα να αναφέρω. Έχουμε το, την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για το Κλίμα, την έκθεση της Greenpeace, της Euro Electric, της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βεβαίως για την Ευρώπη 2050, της ΕΕ για την Οικονομία και, και της Γενικής για την Ενέργεια και της World Wildlife Fund. Μια κύρια παρατήρηση. Η αποδέσμευση από τον άνθρακα σημαίνει ουσιαστικά ε, εξηλεκτρισμό της οικονομίας. Αν κοιτάξουμε λοιπόν τις προοπτικές για το μέλλον, για το 2050 Έχουμε πολύ μεγάλη φάσμα, πάνω από 2.500 τεραουάτ την ώρα, δηλαδή κατανάλωση μια ημέρας σε σημερινά δεδομένα, που θα ε, προβλέπουν ορισμένοι από τους φορείς ως δυνατότητα βελτίωσης αποδοτικότητας της ενέργειας η οποία φαίνεται να αποτελεί το κλειδί για τις μακροπροθέσμες προοπτικές στην ενέργεια σε σχέση με την αποδέσμευση από τον άνθρακα. Εξηλεκτρισμός λοιπόν, electrification στις μεταφορές αλλά και στην θέρμανση, στο τομέα δηλαδή των κτηρίων. Στην προσεχή διαφάνεια θα αναφερθούμε στα πέντε σενάρια για την Ευρώπη, για την αποδέσμευση. Το ένα αφορά την αποτελεσματικότητα στην ενέργεια, έχουμε την διαφοροποιημένη προσφορά, υψηλή περιεκτικότητα σε πυρηνική, χαμηλή περιεκτικότητα σε πυρηνική και ούτω καθεξής. Στην ε, γαλάζια επιφάνεια της διαφάνειάς μας, του σχήματος, βλέπετε τα, όλο φάσμα που καταλαμβάνουν τα πέντε διαφορετικά σενάρια και μετά με τις ε, χρωματιστές γραμμές τα επιμέρους σενάρια. Εντυπωσιακό είναι πάντως ότι ήδη για το 2020 η κατανάλωση ενέργειας με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραμένει λίγο πολύ σταθερή. Δηλαδή πολύ μεγάλη προσοχή δίνεται στην πλήρη ανάπτυξη, τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας. Η γαλάζια γραμμή είναι η αποδοτικότητα της ενέργειας ε, και έχει τεράστια σημασία όπως βλέπετε για τη συνολική κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στο μείγμα δυναμικού που θα μπορούσε να βοηθήσει την Ευρώπη σε στην μετάβαση σε ένα σύστημα αποδέχνωση από τον άνθρακα. Και από τη δική μας θέση βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για το Κλίμα με τη δεύτερη στήλη στη γραφική μας παράσταση, δεύτερη από τα αριστερά, η οποία παρουσιάζει το πιο, η οποία έκθεση το πιο λεπτομέρες σενάριο ως ε, προς τα επίπεδα και το μείγμα που μπορούμε να προβλέψουμε σε ένα από τα σενάρια αυτά. Δηλαδή έχουμε ένα καλό μείγμα με ανανεώσιμες, με θερμική, με φυσικό αέριο και μετά έχουμε βέβαια και την ηλιακή και την αιωλική ενέργεια από την ανοιχτή θάλασσα με πάνω από χίλια Μεγαβάτ τουρμπίνες φυσικού αερίου. 1000 τεραβάτ. Και έτσι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποδεικνύονται να είναι η πιο σημαντική λύση εάν θέλουμε να προχωρήσουμε προς ένα σύστημα αποδεσμευμένο από τον άνθρακα. Ανανεώσιμες λοιπόν πηγές ενέργειας και για λόγους χρονικούς αλλά και για χωρικούς λόγους. Ως προς το χώρο, τα τελευταία χρόνια οι μονάδες παραγωγής ε, βρίσκονταν πάντα στο τόπο κατανάλωσης κοντά. Με την μετάβαση λοιπόν σε αυτές τις νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούμε να έχουμε σύλληψη της ενέργειας σε ένα τοπίο, Φερρυπίν σε ένα χώρο, Φερρυπίν στη Νότια Ευρώπη και μεταφορά της και κατανάλωσή της σε άλλο μέρος, Φερρυπίν τη Βόρεια Ευρώπη. Ανοίγει λοιπόν ε, το φάσμα και το χωρικό αλλά και το χρονικό και βεβαίως με την ε, προοπτική της αξιοποίησης αυτών των ανασωνώσιμων ε, πηγών ενδέχεται και να έχουμε πλεόνασμα ενέργειας, δηλαδή ενέργεια που να μην απορροφάται και να πρέπει να είναι δυνατόν να αποταμιευτεί για μεταγενέστερη χρήση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα τι προβλέπει σε σχέση με τα μείγματα δυναμικού με την διαφάνεια παριθμών 12 όπου εν γέννη διαπιστώνουμε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει επίσης ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, ωστόσο έχει παραλείψει την καταγραφή του δυναμικού που θα χρειαστεί το backup το λεγόμενο για την εξορόπιση του συστήματος μακροπρόθεσμα. Για διάφορους λόγους και περιορισμούς ε, που γνωρίζουμε όλοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πάντως πρέπει να τους έχουμε υπόψη. Για να περάσω στην επόμενη διαφάνεια με το ενεργειακό μείγμα, τον όγκο δηλαδή ενέργεια σε μια αποδεσμευμένη από άνθρακα οικονομία. Οι νέε τεχνολογίε λοιπόν σε όλα τα σενάρια, ακόμα και στο σενάριο ε, high res, παρουσιάζουν κάπου 20% του όλου μείγματο και η πυρηνική ενέργεια και η βιομάζα και το φυσικό αέριο Έχουν λοιπόν ε, σημαντικούς περιορισμούς ως προς τις εκπομπές. Και έτσι φτάνουμε στα κύρια μηνύματα και τις προκλήσεις, ότι δηλαδή μπορούμε με μεγάλο μείγμα, με ευρύ δίκτυο, να προχωρήσουμε αποτελεσματικά προς την αποδέσμευση των άνθρακα. Χωρίς όμως ευρύ δίκτυο ε, δεν μπορούμε και ανανεώσιμες πηγές δεν μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα. Και εδώ μιλούμε βέβαια και για την ε, αποδοχή και για το κόστος, ε, για την εξορροπήση του κόστου στο μέλλον και για το δυναμικό. Όλα αυτά πρέπει να συντηθούν στο δημόσιο διάλογο. Δεύτερο επιχείρημα και μήνυμα. Χρειάζεται ανάπτυξη σε μεγάλο βαθμό των ανανεώσιμων και από το 2030 ήδη αλλά και μετά βέβαια. δεν γνωρίζουμε τι είδους συνέπειες μπορεί να έχουν τα ποσά αυτά στις κοινωνίες μας. Εάν παραδείγματι διανοηθούμε ότι μπορεί να υπάρχουν 600 γιγαβάτ αιωλικής ενέργειας στην ανοιχτή θάλασσα, ενώ στην ε, στεριά πολύ χαμηλότερη παραγωγικότητα, ε, θα συνεπαγόταν αυτό μια ανεμογεννήτρια σχεδόν σε κάθε χωριό, πράγμα το οποίο βέβαια και για λόγου χωροταξίας και προγραμματισμού χωροταξικού δεν μπορεί να ε, κρυθεί αποδοτικό ή και δυνατόν. Γι' αυτό χρειάζεται καλύτερο προγραμματισμό, όπω είπα, αιωλική ενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα, ηλιακή ενέργεια στην Νότια Ευρώπη και αντίστοιχα δυνατότητα μεταφοράς της ενέργειας και αξιοποίησης της και από τη μια πλευρά και από την άλλη. ευελιξία, αξιοποίηση των πόρων και αξιοποίηση των ε, μεγάλων προκλήσεων ε, με ευελιξία που είναι ο τρίτος στόχος, το τρίτο μήνυμα. Καταρχά, σαν πρώτο βήμα με τον περιορισμό του, των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και στη συνέχεια με την ανάπτυξη περισσότερη ε, ενέργεια, αποθήκευση ενέργεια και ενδεχομένω διαθεσή και σε άλλου καταναλωτέ. Και τέταρτον, η πυρηνική ενέργεια, που είναι παρούσα σε κάθε σενάριο. Συνεχίζω ως με την πέμπτη πρόκληση και μήνυμα στο σενάριο που μας μιλάει για βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη χρήση της ενέργειας. Άρα το σενάριο που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, είναι μάλλον δυσβάστατο, δυσβάστατο για τις ε, κοινωνίες και πολύ λίγη δουλειά έχει γίνει ακόμη ως προς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Και εν τέλει θα πρέπει ο επενδυτή να έχει μακροπρόθεσμη ορατότητα, σταθερή και διαρκή ή με κάποια σημαντική διάρκεια ε, εικόνα του νομοθετικού πλαισίου αλλά και του πλέγματος της ενέργειας. Γιατί δεν μπορεί κανείς να κάνει επενδύσεις εκατομμύριων ευρώ εάν δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή η ενέργεια που θα παράγει θα μπορεί να μεταφερθεί και να διατεθεί μέσα από ένα δίκτυο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε μέσα στο λόγο για 10 λεπτά πάλι στον Στέφαν Λέχτενμπερμερ από το Ινστιτούτο Βούπερταλ. Παρακαλώ. Thank you. Uh, dear Mrs. Uh, Sartori, Mrs. Uh, Αγαπητή κυρία Σαρτόρη, κυρία Τζαβέλα, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την πρόσκληση που μου απευθύνετε. Για να μιλήσω εδώ ε, σχετικά με τον ε, ε, ενεργειακό οδικό χάρτη του 2050 βάσει και μιας μελέτης που κάναμε. Στη μελέτη αυτή εμείς, όπως άλλωστε είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, συγκρίναμε διάφορα ε, σενάρια σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Δικό Χάρτη και βλέπετε ε, ότι έχουμε πάλι υπόψη μας την Euroelectric, την Greenpeace και την ECF. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο σύστημα ηλεκτρισμού, γιατί το σύστημα ηλεκτρισμού ε, είναι αυτό το οποίο παίζει κεντρικό ρόλο ε, και στον ενεργειακό δικό χάρτη και στην ίδια την ε, οικονομία που θα είναι απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα. Βλέπετε ότι η μείωση φτάνει στο 99% και βεβαίως το σύστημα έχει μεγάλη διασύνδεση, ε, επομένως υπάρχει και μεγάλος ε, κίνδυνος ε, να φτάσουμε σε αδιέξοδα εάν δεν είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά την μετάβαση από τη μία κατάσταση στην άλλη στον τομέα αυτό. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω κάνοντας κάποιες σύντομες ε, συγκρίσεις. Εδώ είναι οι κύριες στρατιστικές για την απαλλαγή από εκπομπές ε, άνθρακα καθώς επίσης ε, και οι διάφορες δυνατότητες για χρήση πυρηνικών αλλά και εναλλακτικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βλέπετε ότι γενικώ εκτός από το CCS ε, τα υπόλοιπα είναι περίπου συμβατά. Όπως υπόθηκε και προηγουμένως, όλα αυτά βρίσκονται περίπου στο ίδιο επίπεδο με τα προβλεπόμενα από άλλα σενάρια. Θα ήθελα να ασχοληθώ πρώτα με το θέμα της ε, ε, ε, ισχυρής ανάπτυξης στην στην an Η ζήτηση ηλεκτρικού, ε, η οποία θεωρείται ως ε, κοινή στρατηγική σε όλα τα σενάρια. Βλέπουμε ότι μεταξύ του 2005 και του 2050 οι διαφορές έθινε πάρα πολύ μεγάλες όμως ε, στους παραδοσιακούς τομείς χωρίς τον τομέα των μεταφορών. Βλέπουμε ότι τα πράγματα παραμένουν περίπου στο ίδιο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν αυτή την αύξηση που προβλέπουμε Βλέπετε να φτάσει μέχρι το 50% και θα πρέπει οπωσδήποτε ε, να κρατηθεί σε πιο ήπια ε, ποσοστά. Ε, όσον αφορά πάντα την ζήτηση, βλέπουμε εδώ μια διαφάνεια σχετικά με τις μεταφορές και εδώ θα πρέπει να γίνει κάτι έτσι ώστε να υπάρξει μικρότερη ζήτηση όσον αφορά το, τις μεταφορές σε σχέση και με το σύστημα θέρμανσης αυτό ε, είναι ε, ένα ε, σημαντικό σημείο της στρατηγικής όσον αφορά την απαλλαγή εκπομπών άνθρακα και για το ηλεκτρικό σύστημα αλλά και για άλλα. Τώρα, έχει ήδη αναφερθεί, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μελλοντικού σενάριου είναι η μεγάλη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βλέπουμε στην ουσία τρεις ομάδες. Η μία ε, είναι μία περίπτωση με το 1 τρίτο περίπου ε, ε, χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπου είτε δεν έχουν πολλές ανανεώσιμες πηγές είτε χρησιμοποιείται πολύ η πυρηνική ενέργεια. Φτάνουμε στο άλλο τμήμα, υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία φτάνουν ε, στην, ε, στο 80 μέχρι και 98% και στο σενάριο αυτό εμπίπτει και το σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί βέβαια προβλέπονται σημαντικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά την ε, πτυτικότητα του συστήματος και όσον αφορά ε, διαφορετικές, πιο ευέλικτες, ε, μεγαλύτερη ευελιξία και βεβαίως μεγαλύτερη επέκταση και τις δυνατότητες αποθήκευσης και των εφιών κόμπων κτλ. Έχουμε και ένα τρίτο σενάριο που είναι είναι περίπου ανάμεσα από τα δύο. Δύο τρίτα της ε, ε, ηλεκτρικής ενέργειας να έρχεται από ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας και εδώ βεβαίως χρειαζόμαστε ποικιλία και ευελιξία αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε εδώ να χρησιμοποιήσουμε και τη δέσμευση του άνθρακα αλλά και την πυρηνική ενέργεια. Εδώ βλέπουμε κάποια, κάποιες ιδέες που κρύβονται πίσω από τα σενάρια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 πρώτον το ε, κεφαλαιακό κόστος των φωτοβολταϊκών ε, που είναι αρκετά σημαντικό σε σχέση με άλλες ε, τεχνολογίες. Εδώ το συγκρίνουμε. Βλέπουμε επίσης και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ξεκινάει με πάρα πολύ ψηλό κόστος για τα φωτοβολταϊκά αλλά προχωράει με σημαντική μείωση. Η Euroelectric ξεκινάει από πιο χαμηλά αλλά τελικά μειώνεται λιγότερο. Βλέπουμε κι άλλα. Αν δείτε την παρούσα κατάσταση θα δείτε ότι ήδη το 2010 το κόστος ήταν χαμηλότερο από το σενάριο που είχε προβλέψει η ECF. Ε, βλέπουμε εδώ ότι μεταξύ του 2020 και του 2030 επιτυγχάνεται αυτή η καμπή μεγάλη, ε, όμως θα πρέπει να περιμένουμε τις πραγματικές εξελίξεις. Ε, τώρα θα προχωρήσω με κάποια σύντομα συμπεράσματα. Ο ενεργειακός οδικός χάρτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ταυτίζεται και παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με άλλα σενάρια ε, τα οποία ε, αφορούν μελέτες από διάφορους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, ε είναι σημαντικό ε, να έχουμε αποτελέσματα και ε, η πολιτική δράση είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτή την έννοια. κεντρική στρατηγική του οδικού χάρτη του 2050 είναι η απαλλαγή του ηλεκτρισμού από, από τον άνθρακα. για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να, αντιμετωπίσουμε, να το αντιμετωπίσουμε σαν ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί πολυμερώς. Δηλαδή ότι πρώτα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, ενεργειακής ε, ασφάλειας ε, και βεβαίως τα μέτρα όσον αφορά το τμήμα της ε, ε, ζήτησης και της κατανάλωσης στο σύνολό της είναι ε, σημαντικά γιατί πάντα μπορεί να έχουν επίπτωση αντίθετη από αυτή που περιμένουμε. Δεύτερον, στα σενάρια αυτά δεν υπάρχει κανένας χώρος για τα ε, για τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Ε, στην ECF ενδεχομένω ε, γίνεται μια μικρή αναφορά για πολύ λίγες ώρες χρήσης ανά Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οπωσδήποτε θεωρούνται κεντρικό σημείο. Πάντα θα βρίσκουμε μεγάλα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επομένως ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οποιοδήποτε κι αν είναι το σενάριο. Είναι ε, ε, ποικίλε οι και επομένως θα πρέπει να ε, προσαρμόσουμε το σύστημα σε αυτά τα μεγάλα ποσοστά. Όσον αφορά την, το CCS, δέσμευση, αποθήκευση άνδρακα και το πυρηνικό και την πυρηνική ενέργεια, υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες. Νομίζω ότι είναι πολύ χαμηλή η πιθανότητα να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Το πολύ πολύ 30% καθένα. Και αυτό άλλωστε καταδεικνύεται και στις διάφορες μελέτες τις οποίες έχουμε συγκρίνει. Ε, ευχαριστώ πολύ και το σύνολο της παρουσίασής μου μπορείτε να το βρείτε και στο ε, διαδίκτυο. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Λέχτεν Μπέμερ. Έχουμε τώρα λίγο χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Ερωτήσεις μονόλεπτες παρακαλώ έτσι ώστε οι πανελίστες να μπορούν να απαντήσουν. Ε, πρώτη ερώτηση, Βαν Μπρέντ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ τους καλεσμένους μας. Έχω μερικές ερωτήσεις, γιατί και οι δύο μιλήσατε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά οποιοδήποτε μελλοντικού ενεργειακού συστήματος. Τώρα συζητάτε ποιο θα είναι το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών μέχρι το 2050 στο ενεργειακό μείγμα. Μιλήσατε για offshore ενέργεια, onshore, αιωλική και είπατε ότι υπάρχει τεράστιο δυναμικό για παραγωγή ενέργειας χαμηλή, μικρής κλίμακας στις πόλεις, ε, χρήση αιωλικής ενέργειας. Στα δικά σας σενάρια λαμβάνετε υπόψη και αυτό το δυναμικό για αιωλική ενέργεια μικρής κλίμακας, ε, εκμεταλλευόμενη τον ε, άνεμο στις πόλεις για παράδειγμα, αιωλική ενέργεια στις πόλεις. Μιλήσατε και ήδη για το CCS, ε, τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Και είπαμε ότι το φυσικό αέριο θα είναι μια ενεργειακή πηγή που θα μειώσει τη χρήση άνθρακα και θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εμεί ω πολιτικοί θα πρέπει να ιεραρχήσουμε τι προτεραιότητε μα και να δούμε πού θα επενδύουμε στο μέλλον. Και αν θα επενδύσουμε σε δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, δεν θα πρέπει να συνδυάσουμε τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα με το φυσικό αέριο και όχι με τον άνθρακα. Γιατί υπάρχει διαφορά στι τεχνολογίε, Δεν είναι η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιείται ανάλογα με το τι συνδυασμό χρησιμοποιείται. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Χολ. Ευχαριστώ. Κύριε Φωστιέ. Έχω σε εσά μια ερώτηση κυρίως. Είπατε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για τουρμπίνες φυσικού αερίου προκειμένου να εξισορροπηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είπατε όμως ότι μέχρι το 2040 όλα τα ορυκτά καύσιμα θα πρέπει να έχουν σύστημα δέσμευσης αποθήκευσης άνθρακα. Οπότε αν έχουμε στο φυσικό αέριο τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα για να περιορίσει εκπομπέ, ε, δεν έχει την ίδια εξορροπητική δυνατότητα. Πιστεύετε ότι στο μέτρο που προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διασύνδεση, αν θέλουμε μια γνήσια εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από τη στιγμή που θα το κατορθώσουμε, θα μπορούσαμε να ε, το εξισορροπήσουμε, γιατί πάντα θα έχουμε αέρα σε μερικές ε, χώρες και πάντα θα έχουμε ήλιο σε άλλες χώρες και να εξασφαλίσουμε διασύνδεση και αυτού του σενάριου με τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Ευχαριστώ κύριο Ρόιλ. Ευχαριστώ. Έχω καταρχάς την ερώτηση τι σημασία αποδέτε στην πυρηνική ενέργεια στο σενάριο αυτό για το μέλλον εάν θέλουμε να επιτύχουμε σύντομα τους στόχους για το διοξείδιο του άνθρακα. Και δεύτερον, θα ήθελα συγκεκριμένε πληροφορίες για το κατά πόσον έχετε ρεαλιστική εικόνα του κόστους της ωφέλειας από την αποδέσμευση από το διοξείδιο του άνθρακα και την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών, καλά, καθώς και την χρονική, το χρονικό ορίζοντα. Νομίζω ότι είναι λογική ερώτηση. Τι περιμένετε να κοστίσει και πώς θα κρατήσει. Κύριε Δελκαστήγια. Ευχαριστώ. Εγώ έχω μία πιο γενική ερώτηση και ξεκινάει κυρίως από τις υποθέσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που διέπουν και την πρότασή της. Γιατί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μία αλλαγή του μοντέλου στον ενεργειακό τομέα. Και το πιο σημαντικό στην αλλαγή αυτού του μοντέλου είναι ότι η περιβαλλοντική πολιτική και η πολιτική κλιματικών αλλαγών φαίνεται ότι υπερισχύουν ε, της ενεργειακής πολιτικής που φαίνεται ότι εξαφανίζεται από το πολιτικό της πρόγραμμα. Γιατί βασικές ανησυχίες για την ενέργεια, όπως είναι η εξασφάλιση του ενεργειακού ενεφοδιασμού, Η ανταγωνιστικές τιμές, φαίνεται ότι τέτοιου προτεραιότητες επισκιάζονται. Η ενέργεια ε, θα προέρχεται κυρίως από την πυρηνική ενέργεια και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το φυσικό αέριο θα είναι μια μεταβατική πηγή παραχής ενέργειας. Κατά κάποιο τρόπο το ίδιο και, το άνθρακα, ε, και ο άνθρακας τα αυτοκίνητα θα κινούνται με ηλεκτρισμό. Οπότε σε τελική ανάλυση η ενεργειακή πολιτική όπως την φαντάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι περιβαλλοντική πολιτική και πολιτική ε, κλιματικών αλλαγών. Φαίνεται ότι αυτές είναι οι δύο πρωταρχικές ανησυχίες ευρωπαϊκής ε, πολιτικής που πρετανεύουν οποιασδήποτε άλλης. Οπότε ο δικός αυτός χάρτης για την ενέργεια ουσιαστικά είναι ε, χάρτης που επιδιώκει την υλοποίηση περιβαλλοντικών στόχων και κλιματικών αλλαγών. Και φαντάζομαι θα επιδιώξει διεθνή συμφωνία για να υλοποιηθεί, αλλιώς δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Αυτό που ισχύει είναι ότι οι προοπτικές για μια διεθνή συμφωνία για να εφαρμόσουμε ακόμη και αυτό το όραμα της ενεργειακής πολιτικής που θα υπακούει στους στόχους των κλιματικών αλλαγών δεν διαφαίνεται αυτή η προοπτική. Ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν. Η κυρία Ματσέη Κουκ. Ε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα πώς προφέρετε το όνομά μου ότι μου δώσατε το λόγο. Ονομάζομαι Μαζέη. Πάντα υπάρχει πρόβλημα με την προφορά του ονόματός μου. Σας ευχαριστώ πάντως που μου δώσατε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υποβάλω μερικές ερωτήσεις. σε ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη μας ενεργειακή πολιτική. Κατά τη γνώμη μου, αυτή η πολιτική θα πρέπει να είναι ασφαλής και ανεξάρτητη σε μια πρώτη φάση και αργότερα να θέσει και κάποιους περιβαλλοντικούς στόχους, στην περιορισμό δηλαδή της επίδρασης ε, στο περιβάλλον. Έχουμε και το θέμα της ε, θερμότητας, θερμικής ενέργειας. Το 2050 ένα τρίτο της ενέργειας, αν δεν κάνω λάθος, θα προέρχεται από τη θερμική ενέργεια. Και κάτι άλλο. Ποια είναι η στρατηγική λοιπόν ε, που θέλετε να εφαρμόσετε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. σε σχέση με τα υπόλοιπα, με τα κατάλοιπα που αφήνουν. Πώς θα γίνει η διαχείριση αυτών των καταλήπων μέχρι το 2050. Για, τις φωτοβολτα... για τη φωτοβολταϊκή ενέργεια και την ηλιακή ενέργεια. Τι γίνεται με τα κατάλοιπα και τι γίνεται με τους επενδυτές. Όσους λοιπόν θα επενδύσουν στην ανάπτυξη τέτοιων δικτύων. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ δύο ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τις υποθέσεις, τα πορίσματα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον οδικό της χάρτη. Τι γνώμη έχετε για, αυτά, για αυτές τις υποθέσεις, ε, ε, για τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και κυρίως για την υπόθεση που χρησιμοποιείται ότι θα χρειαστεί διεθνή δράση ε, για θέματα κλιματικών αλλαγών. Τι, γίνει όμως, τι θα γίνει όμω αν δεν υπάρξει τέτοια παγκόσμια δράση, τι θα γίνει αν εμεί λάβουμε σήμερα κάποιε αποφάσει και δεν μα ακολουθήσουν οι διεθνεί μα εταίροι. Δεν ε, είναι πιθανό να καταλήξουμε σε διεθνή συμφωνία για τα θέματα αυτά. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση. Ο κύριος Λίχτεμπερμερ είπε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι τόσο αξιόπιστες, ε, δεν είναι προβλέψιμες, είναι πολύ μεταβλητές, γι' αυτό και χρειαζόμαστε ε, ένα αποθεματικό ενέργειας. Βέβαια, σήμερα έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτής της εφεδρικής ενέργειας και τι πολιτικό πλαίσιο χρειαζόμαστε για μια αξιόπιστη, ε, αξιόπιστο ανεφοδιασμό ενέργειας. Θέλουμε ναύσματα και τι χαρακτηριστικά θα πρέπει να έχει η δυναμικότητα της αγοράς. Ο κύριος Οντί. Ευχαριστώ. Ε, για τα θέματα ενέργειας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε φυσικά ε, την επιστήμη, την τεχνολογία και ως προς αυτό το σχέδιο και την πτυχή αυτή και το ΙΤΕΡ, ποια είναι η γνώμη σας, γιατί δυστυχώς ε, ε πριτανεύουν εδώ κάποιες δημοσιονομικές ανησυχίες και όχι επιστημονικές. Το, πιστεύετε ότι το θέμα της σχάσης είναι ε, αξιόπιστο και της πυρηνικής ενέργειας. Για τη γεωθερμική ενέργεια. Εμείς έχουμε ε, γεωθερμική ενέργεια στην πατρίδα μου. Δεν μιλάω για την ε, γεωθερμική ενέργεια επιφάνειας, αλλά βάθους. Μπορούμε εκεί να επενδύσουμε για να εκμεταλλευτούμε τη γεωθερμική ενέργεια. Σε ό,τι αφορά τις υποδομές, τι γίνεται με την πολιτική των υποδομών, σε ό,τι αφορά την ιδιοκτησία των υποδομών. Γιατί σήμερα έχουμε εκατοντάδες διαφορετικούς ιδιοκτήτες ε, ενέργειας ε, ψηφιακής. Ε, μήπως όμως δημιουργήσουμε τεράστιες θεατρικές δημόσιες και εκεί θα έχουμε μια προσπάθεια να συντονίσουμε τις επενδύσεις μας στις επενδύσεις αυτές. Ευχαριστώ κύριος Γκέρεκ. Ευχαριστώ. Φυσικά προσωμιώσεις και προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για τα πάντα. Ιδιαίτερα όταν έχουμε ένα τόσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα όπως το 2050. Αλλά αυτό μου θυμίζει λίγο επιστημονική φαντασία. Γιατί δεν έχουμε προσωμιώσεις που θα λαμβάνουν υπόψη όλους τους πολιτικούς στόχους. Το στόχο της ασφάλειας, τον κλιματικό στόχο, το στόχο των εκπομπών. Η λύση βρίσκεται κάπου στη χρυσή τομή, αλλά δεν έχουμε κάποια προσωμείωση για την βελτιστοποίηση. Γι' αυτό και έχω μία ερώτηση. Ε, έχουμε ε, εργοστάσια ε, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση άνθρακα. Το διαγράφεται όμως, χρησιμοποιείται περισσότερο το CCS, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Δεν υπάρχουν όμως αρκετές έρευνες για το CCS. Συνεχίζονται οι δοκιμές και τα πειράματα. Δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ηλεκτρικού σταθμού ε, που θα χρησιμοποιεί άνθρακα μεν, αλλά καθαρό άνθρακα. Κάποτε μιλήσαμε και αυτό το καθαρό άνθρακα, το clean coal, με αποτελεσματικότητα 50%. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 20-30 χρόνια τέτοιου, έχουμε 20-30 χρόνια μπροστά μας μέχρι το 2050 για να δημιουργήσουμε τέτοιες, ε, τέτοια εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με χρήση καθαρού άνθρακα. Τι γνώμη έχετε για αυτή την πιθανότητα. Η κυρία Έρτσοκ. Ευχαριστώ και να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, να ρωτήσω τον κύριο Στέφαν Λέχτενμπέμερ αν ασχολήθηκε καθόλου με τον περιφερειακό αντίκτυπο, γιατί δεν υπάρχει ομοιογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα κράτη-μέλη στο μέλλον θα πρέπει να κάνουν τις δικές τους επιλογές ε, ανάλογα με τις πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να δούμε και την περιφερειακή πηγή. Δεν υπάρχει ομοιόμορφη αγορά ενέργειας αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Με αυτό το θέμα το περιφερειακό ασχοληθήκατε. Και από την GDF Suez ε, θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο. Όλα αυτά τα ενεργειακά προγράμματα ε, δημιουργούν τεράστιες ευθύνες γιατί θέλουμε να διπλασιάσουμε την παραγωγή ενέργειας και ταυτόχρονα λάβουμε υπόψη και το περιβάλλον και να επενδύσουμε στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών. Οι επενδύσει για το περιβάλλον είναι πιο ομοιόμορφε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ στην ενέργεια έχουμε πολύ διαφορετικές, ε, διαφορετικά επίπεδα και προκλήσει. Χρειαζόμαστε επενδύσεις και για τις νέες ε, εγκαταστάσεις, αλλά και για τον καθαρισμό των, των υπαρχουσών εγκαταστάσεων. Χρειαζόμαστε λοιπόν για την ενέργεια φαινό επενδύσει, αλλά χρειαζόμαστε επενδύσεις και για το περιβάλλον, για τις κλιματικές αλλαγές. Αυτές οι επενδύσει στην Ευρώπη πώ ε, δρομολογούνται κατά τη γνώμη σας. Ευχαριστώ κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Έχουμε κάποιους στόχους, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να δούμε με ποιε μεθόδους και ποιου τρόπους θα υλοποιήσουμε αυτού του στόχου. Γιατί θα πρέπει να χαράξουμε και τη μέθοδο για την υλοποίηση αυτών των στόχων γιατί ζούμε μια κρίση, υπάρχει αυτή η κρίση ε, και θα κρατήσει ακόμη. Τι δημοσιονομικά κονδύλια προβλέπουμε για αυτούς τους στόχους, λοιπόν, να εξέλθουμε από την κρίση και να υλοποιήσουμε τους στόχους. Έχουμε και την Ευρώπη 2020 και πέρα από το 2020. Όλοι αυτοί οι στόχοι φαίνεται ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθούν μέχρι το 2050, δεδομένου ότι κάποιες ευρωπαϊκές οικονομίες στηρίζονται αποκλειστικά στον άνθρακα και μια τέτοια επανάσταση ενεργειακοκλιματική, περιβαλλοντική θα είναι αδύνατη, ανέφικτη σε ορισμένες περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκαν οι ε, ερωτήσεις και θα δώσουμε ε, στον κάθε ομιλητή τρία λεπτά έτσι ώστε να δώσει κάποιες γενικές απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω μια σύνοψη των ερωτήσεων έτσι ώστε να απαντήσω συνολικά. Ε, η ερώτηση η οποία επανέρχεται αφορούσε την τεχνολογία. Αυτές ε, είναι εξωτερικές απόψεις. Πώς όμως μπορούμε, πώς μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις ε, ε, μελέτες αυτές. Ναι, είναι γεγονός ότι χρειαζόμαστε όριμες τεχνολογίες. Ε, οι θαλάσσιες τεχνολογίες ας πούμε δεν έχουν συνυπολογιστεί ή πολύ λίγο. Και για να επανέλθω και στην ερώτησή σας ε, κυρία Βαν Μπρέντ, ε, μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ναι όσον αφορά τον ήλιο, όσον αφορά τον αέρα, ε, είναι τελείως διαφορετικά αν μιλάμε για γεννήτριες ή onshore ή offshore ε, ή αν μιλάμε για μεγάλες ε, μονάδες που μπορούν μαζικά να δημιουργήσουν ανανεώσιμη ενέργεια. αλλά εάν αυτές οι μεγάλες περιοχές, οι επικεντρωμένες λειτουργήσουν. Ναι, ίσως πρέπει να πάμε σε μικρές, ε, ενέργειες, σε μικρές μονάδες ε, για τη γεωθερμία. Ναι, δεν έχει συνυπολογιστεί. Ε, μακροπρόθεσμα πάντως φαντάζομαι ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν τμήμα του ενεργειακού μείγματος. Στο μέλλον όμως. 500.000 ε, ΜΒ που αναφέρονται στη μελέτη ECF συγκρινόμενα ε, με την μαζική αντικατάσταση των συνδέσμων, των grids, τα εφηή δίκτυα ε, είναι ε, γεγονός ότι είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι δυνατόν μέσω ε, διεύρυνσης του εφιούς δικτύου να αναπληρώσει κανείς τις άλλες λήψεις και φέτος το χειμώνα στην Ευρώπη Είχαμε, είχαμε ένα πρόβλημα ε, γιατί είδαμε ότι πολλές ε, χώρες ακόμα βασίζονται στο ηλεκτρικό και επομένως κάποια στιγμή ε, υπήρξε ανάγκη για μαζική παραγωγή. Ο μελλοντικός ρόλος του CCS, δέσμευση αποθήκευσης άνθρακα για το άνθρακα και για το αέριο δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ποσοστό του καθενός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε ένα σύστημα που δεν θα υπάρχει, δεν θα προβλέπεται καθόλου η πυρηνική ενέργεια ή το CCS είτε αφορά τον άνθρακα είτε αφορά το φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να έχουμε μείγμα χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτά. Yes, I will try. Θα προσπαθήσω και εγώ να απαντήσω τις ερωτήσεις οι οποίες αφορούν την τεχνολογία. Το θέμα του CCS βεβαίως είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν και άλλα ερωτηματικά όσον αφορά το CCS. Αυτή τη στιγμή τα ερωτηματικά είναι περισσότερα από τις ε, απαντήσεις. Η τεχνολογία θα πρέπει να δώσει απαντήσεις. Τώρα όσον αφορά την ε, σχέση του άνθρακα και του φυσικού αερίου σε σχέση ε, και με την κλιματική αλλαγή είναι η δυνατότητα αποθήκευσης ε, είναι ε, πολύ σημαντική και βεβαίως θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο φυσικό αέριο. Υπήρξε και μια άλλη ερώτηση σχετικά με την κλιματική πολιτική. Τα προβλήματα του κλίματος δυστυχώς θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν και επομένως πολλές από τις πολιτικές πολιτικές και τα σενάρια θα πρέπει να είναι καλά και όσον αφορά την προσφορά και όσον αφορά τις ενέργειες ε, και την ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και όσον αφορά και άλλα θέματα. Ε, τώρα ε, ο άνθρακας βεβαίως είναι πρόβλημα όσον αφορά το περιβάλλον αλλά ε, πρέπει να πούμε ότι ακόμα και το πράσινο, το πιο οικολογικό ε, κάρβουνο, ε, ο πιο οικολογικός άνθρακας, και αυτός παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λαμβάνει υπόψη της το θέμα αυτό εμείς ε, σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο ε, πρέπει να ληφθεί υπόψη, πρέπει να καλυφθεί και αυτό το ζήτημα και οπωσδήποτε να, ληφθεί καλύτερα, να ληφθούν καλύτερα υπόψη, μάλλον οι διαφορές που παρουσιάζουν διάφορες περιφέρειες. Όσον αφορά τώρα τα οικονομικά ζητήματα, προσωπικά πιστεύω ότι έχουμε πολλές ε, πιθανότητες επιτυχίας με την επένδυση αλλάζουμε πολύ το σύστημα. Απομακρυνόμαστε από το ισχύον, το παλιό σύστημα, πάμε προς νέα συστήματα. Και ε, κατά αυτή την έννοια μπορούν να δημιουργηθούν πολλές ε, ε, ευκαιρίες για ανάπτυξη, για δημιουργία θέσεων εργασίας θεωρώ ότι αυτό είναι από τους πιο ενδιαφέρουσες, ενδιαφέροντες τομείς που μπορούν να βοηθήσουν την υπέρβαση των προβλημάτων, την υπέρβαση κρίσεων ε, και βεβαίως ε, θα πρέπει να βρούμε και τις δυνατότητες ιδιωτικής χρηματοδότησης για τους τομείς αυτούς. Ε, είναι μεγάλες οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας αλλά και πολλά υποσχόμενες. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ τους ε, εισηγητές μας ε, που με πολύ συνθετικό τρόπο κατάφεραν να απαντήσουν. Θα πρέπει να αλλάξει φρουρά τώρα. Μέχρι να καθίσουν οι άλλοι εισηγητές ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. και πρέπει να σας πω ότι την επόμενη φορά που θα οργανώσουμε κάτι τέτοιο δεν θα δεχτώ έξι ομιλητές. Ναι, τέσσερι το πολύ, έξι δεν είναι δυνατόν, γιατί διαφορετικά θα είμαστε πάντα σε αυτή την κατάσταση, τρομερά αργοπορημένοι. Ξέρετε ότι έχουμε ακόμα τέσσερι εισηγήσει να ακούσουμε, γι' αυτό σα παρακαλώ όταν θα πάρετε το λόγο ε, να, είμαστε, να σεβαστείτε το χρόνο, τουλάχιστον να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μιλήσουν, να τους ακούσουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω αμέσως το λόγο για το δεύτερο σκέλος της συνάντησής στον κύριο Χάβαρτ Βάγγεν Μάλβικ από την Statcraft AS. Κύριε Μάλβικ, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. θα προσπαθήσω να τα πω λίγο πιο γρήγορα για να προλάβω. Εκπροσωπώ την Stratcraft, την ε, νορβηγική εταιρεία. Με παγκόσμιο εμφέλιο που παράγει την, ε, τις ανανεώσιμες ποιες ενέργειας της Ευρώπης στο ποσοστό. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό μας. Αυτό θα αναφερθώ λοιπόν στην κατάσταση στην Ευρώπη από τη δική μας οπτική γωνία και για τα επόμενα χρόνια. Όπως γνωρίζετε τώρα, έχουμε εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εγκαταστάσεις για την ανανόσιμη ενέργεια που πηγαίνουν καλά. Πράγμα το ικανοποιητικό μεν, υπάρχουν όμως και κάποιες άλλε εξελίξεις. Οι τιμέ του άνθρακα και το σύστημα των ανταλλαγών δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Δεν έχει φέρει αποτελέσματα η τιμή και μεταστροφή στην αγορά από τον άνθρακα προς το φυσικό αέριο λόγω των πολύ χαμηλών τιμών. Αυτό είναι το ένα πράγμα που πρέπει να έχουμε υπόψη. Και δεύτερον, η ενέργεια που διατηρείται στην Ευρώπη είναι πάγια λίγο πολύ και δεν θα μεταβληθεί στα επόμενα χρόνια. Έχουμε δώσει κάποιες ε, απεικονίσεις για την Ευρώπη των 27 και για τη Γερμανία ιδιαίτερως. Ωστόσο αυτό το φαινόμενο προξενεί δυσκολίες και για τους επενδυτές και για τις εταιρείε και λόγω βέβαια της τιμής του άνθρακα και της σταθερής ζήτησης που δεν επιτρέπουν περισσότερες επενδύσεις. Εάν γίνουν προς επενδύσει ανανεώσιμε, τότε ενδέχεται να μειωθούν σημαντικά οι τιμέ αυτών και έτσι θα είναι δύσκολο για μας να προβούμε τι επενδύσει. Δεν θα είναι αποδοτικέ δηλαδή οι επενδύσει μα στι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στην Ευρώπη. Γι' αυτό τίνουμε προ τι άλλε αγορέ έξω από την Ευρώπη. Μια επιλογή στην πολιτική μας. Έχουμε ξανασυστήσει τα θέματα αυτά και στο παρελθόν. Όλες οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας που έχουν κατασκευαστεί άνω την Ευρώπη πρέπει να περάσουν πλέον στον χώρο τη κατανάλωση, Δηλαδή χρειάζεται μαζική ανάπτυξη του δικτύου στα επόμενα χρόνια. Και επίσης δεν υπάρχει να δημιουργηθεί πραγματική ενιαία αγορά ενέργειας εάν δεν βελτιωθεί σημαντικά η διασύνδεση μέσα στο δίκτυο. Βελτίωση λοιπόν του δικτύου και κόστος και αποτελεσματικότητα. Κόστος και απόδοση. Ωστόσο πρέπει να διερωτηθούμε και τι άλλες δυνατότητες, μάλλον ανάγκες υπάρχουν για υποδομές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ακόμη συζητηθεί στην Ευρώπη. Πρέπει να το καλύψουμε ωστόσο. Και για το σύστημα σύλληψης και αποθήκευσης άνθρακα, τι θα γίνει και θα επαναληφθώ σε αυτό αργότερα. Ας δούμε όμως τώρα. Γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε. Ότι αυτά που συζητούμε σήμερα είναι πολύ σοβαρά. Γιατί έχουμε φτάσει σε έξι σε προβολή αύξησης της θερμοκρασίας της γης κατά 6 με 8 βαθμούς. Άρα θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στις προβολές μας. Και ξέρουμε ότι η λίθινη εποχή δεν σταμάτησε λόγω απουσίας λίθων πέτρας, όπως και η εποχή του καυσίμου δεν πρόκειται να λήξει λόγω απουσίας καυσίμου. Καύσιμο θα υπάρχει ακόμη και πετρέλαιο και φυσικό αέριο και άνθρακα στο μέλλον. Χρειάζονται όμως θαραλέες πολιτικές και επιλογές για να μπορέσουμε να βρούμε άλλες λύσεις. Και επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε τη μακροπρόθεσμη δέσμευση για το μέλλον από, τις, από τα ορικά τα καύσιμα, στα ορυκτά καύσιμα, την εξάρτηση δηλαδή από τα ορικά καύσιμα, που θα μας δεσμεύσει σε ένα σύστημα για ακόμη μια 40 ετία, 50 με το σύστημα σύλληψης και αποθήκευσης άνθρακα. Και βέβαια εδώ βλέπουμε ότι μπορεί αυτό να αποτελέσει μια προοπτική. Τα ορυκτά μπορούν να αποτελέσουν ακόμη προοπτική για την επόμενη δεκαετία, αλλά πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο και να τυπωθούν τα ερωτήματα για το κόστος του συστήματος σύλληψης και αποθήκευσης άνθρακα. Τι χρειάζεται να κάνουμε λοιπόν. Ασφαλώς πρέπει να συνεχιστούν ε, να αναπτύσσονται οι πηγές για ε, να στην Ευρώπη. Να συνεχιστεί δηλαδή η θετική στάση προς την βιομηχανία των ανανεώσιμων. Πρέπει να συνεχιστεί η επιδότηση, οι επιδοτήσεις προς την βιομηχανία των ανανεώσιμων για τα επόμενα χρόνια μέσω πρόθεσμα. Αλλά βέβαια μάκρο πρόθεσμα θα πρέπει να είναι και ανταγωνιστικές αυτές οι επιχειρήσεις. Κάποιες έχουν ήδη κάνει προβολές ως το 2020 για την ολική ενέργεια στην ανοιχτή θάλασσα και ίσως εκεί μπορούμε να δώσουμε και με ένα μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο. Χρειάζεται λοιπόν, όπως έλεγα και νωρίτερα, επενδύσεις και στο χώρο των δικτύων και στο χώρο της διασύνδεσης των κόμβων Και αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που διαβλέπουμε για το μέλλον. Θα προχωρήσει ο εξηλεκτρισμός και μια λύση ε, χωρίς ψωγυρίσματα για καλύτερες κλιματολογικές συνθήκες. Χρειάζονται όμως πάνω απ' όλα υψηλές τιμές στον άνθρακα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το ορίσουν μεταξύ άλλων και οι αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιανουάριο, άνωθεν δηλαδή πρέπει να προσδοριστούν αυτές οι τιμές, πρόθεσμα τουλάχιστον, μετά το 2020 όμως μακροπρόθεσμα, θα χρειαστεί ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη διαφορών στην αγορά και την παραγωγή ενέργειας η οποία θα τίνει περισσότερο προς τις ανανεώσιμες λύσεις. Και με μια γελιογραφία που βλέπετε εδώ στα δεξιά κλείνω Μπορεί να λέμε ότι είμαστε καταδικασμένοι εάν προχωρήσουμε σε διαφορετικές λύσεις, αλλά είμαστε πιο πολύ καταδικασμένοι ακόμη εάν δεν προχωρήσουμε. Θα δώσω τώρα το λόγο ε, στον καθηγητή Φέλιξ Χέφνερ από το Ινστιτούτο Ενεργειακής Οικονομίας. Ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να πω λίγα λόγια για τις ευκαιρίες που μας δίνει η μια ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας δώσω δύο παραδείγματα από τον τομέα του ηλεκτρισμού. Το πρώτο αφορά τη δημιουργία δικτύου για την εναρμόνιση τη δυνατότητα εναρμόνισης υποστήριξης των συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δεύτερο θέμα είναι η ασφάλεια του, του ανεφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια και μηχανισμοί δυναμικότητες. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια θα είναι τα πιθανά ωφέλη που θα έχουμε από μια ολοκλήρωση της ε, ενεργειακής αγοράς, ποια είναι τα εμπόδια, τι θα πρέπει να ε, κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπερβούμε αυτά τα εμπόδια και τι να αφήσουμε στα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση τώρα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Συντήρηξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έχουμε το αρμόδιο Ινστιτούτο που ήδη το 2010 έκανε στην Κολονία ε, μία μελέτη για τα ωφέλη της εναρμόνισης ε, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των στόχων για το 2000, της Ευρώπης 2020. Και έχουμε ε, ένα πλεόνασμα κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εναρμόνιση. Και τα ωφέλη της εναρμόνισης απορρέουν, όπως μας δείχνει και η γραφική επικόνηση είναι στο ότι ε, η πιο φθηνέ περιοχές παραγωγή ε, είναι στι εξωτερικέ περιφέρειες Ευρώπη, ε, φωτοβολταϊκά στο νότο, αεολική ενέργεια στο βορρά. Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τι καλύτερε περιοχέ ε, και τον καλύτερο μέθοδο ενέργεια και μετά με το δίκτυο να τι διασυνδέσουμε. Και είναι εύκολο να έχουμε αιωλική ενέργεια στην Ισπανία και να διοχετεύουμε την ενέργεια στη Γερμανία. Είναι πολύ πιο φθηνό από ότι να επιδιώξουμε την αιωλική ενέργεια στην Γερμανία. Τώρα, ποιε είναι οι προκλήσεις. Θα πρέπει να κατασκευάσουμε δίκτυα, όχι μόνο για τους στόχους της Ευρώπης 2020, αλλά και τους στόχους του 2050. Και φαίνεται στο σκούρο χρώμα μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική το 2050. Ποιο είναι το, κόστος, το σενάριο του χαμηλότερου κόστους. Και πάλι στις εξωτερικές περιοχές έχουμε ε, τον ηλεκτρισμό με αιωλική ενέργεια και με αιωλική και φυσικά χρειαζόμαστε μαζική επέκταση αυτού του δικτύου. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο σημείο. Ένα σημαντικό εμπόδιο είναι ε, τι γίνεται με τη διανομή, κάποια προβλήματα διανομής. Έχω εδώ στη μικρή εικόνα το παράδειγμα της Ιταλίας. Η Ιταλία βλέπετε ότι δεν είναι ούτε με σκούρο χρώμα, ούτε ανοιχτό γκρι, αλλά είναι κάπου στη μέση. Οπότε με βάση αυτή την μακροπρόθεσμη προσωμείωση και κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί μέχρι το 2050, πάντως με αυτό το σενάριο η Ιταλία είναι, έχει σε ό,τι αφορά την, τον ηλεκτρισμό, αλλά για να υλοποιηθεί αυτό το σενάριο θα πρέπει να έχουμε μαζική επέκταση δικτύου στην Ιταλία για τη μεταβίβαση ηλεκτρισμού από το νότο, από το νότο προς το κέντρο της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε λοιπόν υψηλό δίκτυο για τη μεταφορά ενέργειας στην Ιταλία. Ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Και εδώ θα πρέπει ε, να καταπολεμήσουμε τις αντιστάσεις, γιατί σε εθνικό επίπεδο δεν χρειάζεται ένα τέτοιο δίκτυο ηλεκτρισμού. Γι' αυτό και χρειάζεται εδώ δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε τι θα πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και την αφήσουμε σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το πιο σημαντικό είναι να έχουμε μία, ένα σαφή στόχο πολιτικής. Αν έχουμε κλιματική πολιτική, σαφείς στόχους και μέτρα για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Να έχουμε μηχανισμούς ε, ομοιόμορφους, ε, ε, ουδέτερους από τεχνολογική άποψη για να βελτιώσουμε την παραγωγή ηλεκτρισμού. Επίση, για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, θα πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό αντισταθμίση, για αυτού που θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν περισσότερο το μηχανισμό από αυτού που θα έχουν πιο άμεσα ωφέλη. Και μία ανακατανομή των κονδυλίων από το κεντρικό προπολογισμό προ τα κράτη-μέλη, δημιουργώντα κάποιου μηχανισμού που θα δίνουν και ενάψματα στους ιδιώτε επενδυτέ για να συμμετέχουν. Και αυτό είναι αρκετά δύσκολο θέμα και θα πρέπει να είμαστε πιο ευρηματικοί στις προτάσεις. Τώρα, σε επίπεδο κρατών μελών, το πιο σημαντικό είναι να εφαρμοστούν οι μηχανισμοί που καταρτίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μην έχουμε επιπλέον συμπληρωματικά εθνικά μέτρα που θα δημιουργούν προβλήματα στη διαμόρφωση τιμής άνθρακα, για παράδειγμα. Δεύτερο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ε, το backup capacity. Χρειαζόμαστε και τέτοιο εφεδρικό δυναμικό να ε, δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση που έχουμε υψηλή ζήτηση ηλεκτρισμού και ε, λιγότερη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε εχμές κυρίως το απόγευμα ζήτησης. Οπότε να μην ε, έχουμε σύμπτωση της ε, αιχμής της ζήτησης με την πτώση του ανέμου και τη χαμηλή παραγωγή. Από πέρυσι τον Νοέμβριο έχουμε κάποια στοιχεία στη Γερμανία. Είχαμε τρει διαδοχικέ μέρε που είχαμε πλήρη άπνοια στη Γερμανία. Και αν ε, σκεφτεί κανεί ότι έχουμε ένα σύστημα παραγωγή ηλεκτρισμού με 40-50% μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βλέπετε τι πρόβλημα είχαμε και πόσα εφεδρική ενέργεια χρειαζόμαστε για να καλύψουμε τέτοιου είδου κενά. Αναφέρθηκε όμως και στη συζήτηση σήμερα εδώ, ότι αν έχουμε πιο ευρωπαϊκή προοπτική και όχι εθνική, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα, την ευρωπαϊκή πολιτική για να μειώσουμε τα προβλήματα από, την, από το εφεδρικό δυναμικό που, που χρειαζόμαστε. Γιατί ε, σε πέντε χρόνια είχαμε μόνο σε μία ώρα αυτή την κατάσταση στη Βόρεια Ευρώπη. Υπάρχει ε, μία διατα... Ε, μία... ένα δυναμικό για ε, τεράστιο χαρτοφυλάκιο, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα αυτό το τα ωφέλη από αυτό το γενικό φεδρικό και να χρησιμοποιήσουμε ε, τέτοιο εφεδρικό δυναμικό για να εξασφαλίσουμε ε, τον ενεργειακό μας ανεφοδιασμό στην ενέργεια. Πάντως χρειαζόμαστε τέτοιο backup capacity εφεδρική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα ολοκληρωμένο δίκτυο, διασυνδεδεμένο, για να υλοποιήσουμε τους στόχους του 2050. Και ένα τέτοιο ε, ανάμεικτο δίκτυο θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη θα εκμεταλλεύονται ε, την ε, ενέργεια που υπάρχει σε άλλα κράτη. Αυτό ίσως δημιουργήσει ενδεχομένως πρόβλημα. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, για παράδειγμα ρύθμιση στο φυσικό αέριο. Και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αποφύγουμε το πρόβλημα του free riding ορισμένων κρατών μέλων εις βάρος ε, άλλων κρατών μέλων. Σε ό,τι αφορά το εθνικό επίπεδο, χρειαζόμαστε λιγότερη εναρμόνιση, γιατί καλή εναρμόνιση, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο καλύπτουν τα θέματα ενεργειακού ανεφοδιασμού τα κράτη-μέλη, όχι μόνο το επίπεδο. Γιατί χρειαζόμαστε κάποιους μηχανισμούς δυναμικού, εμ, πληρωμές, ενιαία αγορά και βλέπουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη κάνουν κάτι, αλλά ο καθένας κάτι, κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά αυτό στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργεί πρόβλημα. Και τέλος, αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο να χρηματοδοτήσει κάτι, ούτε συγκεκριμένες τεχνολογίες ή εταιρείε, αλλά να βρει τους κατάλληλους μηχανισμούς, τους κατάλληλους κανόνες για να δίνει ενάψματα σε ιδιώτες προκειμένου να υλοποιούν αυτούς τους στόχους των πολιτικών. Έτσι θα έχουμε τη μεγαλύτερη ευκαιρία να υλοποιήσουμε τους στόχου της πολιτικής και μάλιστα με το φθηνότερο δυνατό τρόπο. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο οι μηχανισμοί, οι ρυθμίσει και όχι τόσο τα χρήματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για το όσα μας είπατε. Ξεκινάει η συζήτηση. Παρακαλώ πολύ ερωτήσεις να μην υπερβάλλουν τα το ένα λεπτό, συγγνώμη, το ένα λεπτό. Η κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Mr. Malvik, you were very... Κύριε Μάλβικ, διέκρινα μεγάλο σκεπτικισμό όσον αφορά την ε, ανάγκη υποδομής ε, σε ε, υποδομές για το φυσικό αέριο. Είσαστε τόσο βέβαιος ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να δώσουν, να προμηθεύσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μήπως έχετε ε, μόνο κάποια ε, μέλη στην, στο μυαλό σας. Είναι δυνατόν χωρίς φυσικό αέριο γιατί υπάρχουν χώρες που δεν έχουν ούτε έντονο αέρα, ούτε ε, ηλιοφάνεια. Πώς θα επιβιώσουν οι χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ, Βαν Μπρέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τους ομιλητές για τις παρουσίες τους, ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ήθελα απλώ να ενσωματώσω την κοινωνική διάσταση στη συζήτηση αυτή και κυρίω στον τομέα των νόσιμων πηγών, δεδομένου ότι συμφωνούμε όλοι ότι θα αποτελέσουν την ραχοκοκαλιά στη οποιαδήποτε μελλοντική ενεργειακή πολιτική μα. Ε, στην πατρίδα μου, αλλά έχω υπόψη μου και άλλα κράτη-μέλη. Ένα κύριο μέλημα είναι ότι η αύξηση στα τιμολόγια της ενέργειας για τον καταναλωτή οφείλεται στο ότι έχουν γίνει τόσο σημαντικές επενδύσεις στις ανανεωνόσιμες πηγές από τους ενεργειακούς φορείς. Βραχυπρόθεσμα ίσως να εξηγείται αυτό. Αλλά ταυτόχρονα κάποιο άρθρο που διάβασα προσφάτα για τη Γερμανία μας λέει ότι είναι μια από τις πρωτοπόρους στην, ε, στις πηγέ πηγές η Γερμανία στην Ευρώπη τώρα. Με αποτέλεσμα τώρα να αρχίσει να μειώνεται η, η τιμή στην ενέργεια. Ερωτώ λοιπόν στους ομιλητές μας, περιμένουν να συμβεί κάτι, κάτι τέτοιο μεσοπρόθεσμα. Θα αρχίσει να μειώνεται εάν αλλάξει το μείγμα και έχουμε 30, 40, 50, 60% ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μας μείγμα. Θα έχουμε το δυναμικό να μειώσουμε, δεδομένου ότι θα χρειαστούμε και περισσότερες επενδύσεις, ε, να μειώσουμε τις ε, τιμές για τον καταναλωτή στην Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Χολ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα δύο πράγματα να ρωτήσω σχετικά με την εναρμόνιση των προγραμμάτων υποστήριξη. Και πρώτον, γιατί θεωρείτε ότι ποιος είναι ο λόγος την άποψη που δεν έχουν αξιοποιήσει τα κράτη-μέλη τους μηχανισμούς από την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές που πιστεύω θα ήταν και ο απλούστερος αλλά και πιο άμεσος τρόπος να προχωρήσουν στον δρόμο αυτόν. Και δεύτερον, γιατί βέβαια είναι αρκετά ελκυστική η λύση γιατί μειώνονται μειώνεται και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι για να περάσουμε το να περάσουμε ε, συνολικά στην πιο ελκυστική αυτή ε, φάση, ως, η περιοχή καλύτερα ως προς τις ε, ανανεώσιμες πηγές στην πιο ανεμοδαρμένη περιοχή δεν θα έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ ψηλό κόστος και επιπλέον πολύ μεγαλύτερο κόστος σε δίκτυο, σε διαδικτύωση. Ευχαριστώ Χέρτσοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να τον πρώτο μιλητή σε αυτό που ανέφερε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση στις, ε, στη ζήτηση για τα επόμενα χρόνια. οι προηγούμενοι ομιλητέ από το πρώτο πάνελ μα μίλησαν για διπλασιασμό τη ζήτηση. Εάν έχουμε τόσο μεγάλε αποκλήσει λοιπόν απόψε, πρέπει να τι συστήσουμε διεξοδικά. Και δεύτερον, για την ε, δωρεάν εκμετάλλευση των συστημάτων ε, ορισμένων κρατών από κάποια άλλα που αναφέρατε νωρίτερα, το free riding δηλαδή. Υπάρχει όντω αυτή η προοπτική, αλλά υπάρχουν και χώρε οι οποίε διστάζουν να, ε, να βλέπουν την αξιοποίηση κάποιων κοινοτικών κονδυλίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση από ορισμένα κράτη. Άλλου τύπου free riding είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε γενικότερα το φαινόμενο της εκμετάλλευσης των πόρων από ορισμένου μόνο. Για δε το ζήτημα των εξωτερικών, ε, της εξωτερικής ε, προοπτικής για την ενέργεια που είχα εγώ την εισήγηση, διαπίστωσα ότι ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στα, στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά. Ευχαριστώ πολύ. Δύο λεπτά στον κάθε εισηγητή για την απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Uh, um, Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά τους αγωγούς πετρελαίου και αερίου στην Ευρώπη. Θα πρέπει να δούμε τι διαφορές υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών στην Ευρώπη. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα της ζήτησης ε, ενέργειας και ηλεκτρισμού και πόσο θα χρειαστούμε, τι ενέργεια θα χρειαστούμε στο μέλλον. Τώρα μιλούμε για ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα το 2050 και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες δεκαετίες η ζήτηση πριν ε, ε, προτείνουμε τη μαζική κατασκευή υποδομών που θα εγκλωβίσει ουσιαστικά την ενέργεια που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στην Ευρώπη, θα, χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τις επόμενες τρεις-τέσσερις δεκαετίες. Σήμερα πρέπει να γίνει συζήτηση. Απάντηση δεν έχουμε ακόμη. Τώρα, το θέμα της ζήτησης και πάλι σίγουρα δεν θα αυξηθεί. Κατά τη γνώμη μας θα παραμείνει σταθερή η ζήτηση την επόμενη δεκαετία. Βέβαια, αν λάβουμε κάποιες αποφάσεις πολιτικής και ε, δώσουμε έμφαση στον εξηλεκτρισμό διαφορών τομέων, την παραγωγή θερμότητας, ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τότε όντως θα αυξηθεί η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια ανάλογα με τις επιλογές πολιτική. Το θέμα είναι αυτό θα γίνει από μόνο του ή θα πρέπει εμείς να λάβουμε κάποιες αποφάσεις πολιτική για να το πραγματοποιήσουμε. Γιατί ε, ίσως θα πρέπει έτσι να προβλέψουμε και περισσότερο χώρο, μεγαλύτερο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Τώρα, για του τους του ηλεκτρικού. Η απάντηση είναι ότι αν έχουμε μαζικές κατασκευές υποδομών ε, για το δίκτυο, αυτό θα είναι επωφελές και για τους καταναλωτές στην Ευρώπη. Και αν κάθε χώρα μόνη της θα πρέπει να φροντίσει για την ενέργεια, τότε και οι λογαριασμοί θα πρέπει να είναι πιο υψηλοί. Η διασυνοριακή, το διασυνοριακό εμπόριο θα αποβεί προς όφελος και του καταναλωτή, κατά τη γνώμη μου, και των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω και εγώ λίγα λόγια. Σίγουρα ήδη η Ευρώπη έχει ένα ισχυρό μηχανισμό εναρμόνισης, το σύστημα εμπορίας εκπομπών. Το θέμα είναι τι άλλα εργαλεία χρειάζεται και τι άλλους μηχανισμούς θα χρειαστεί για να υλοποιήσει και τους στόχους στο περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Το θέμα είναι θα πρέπει ε, να συνδέουμε τι πιο, αποτελεσ... τις πιο αποτελεσματικές περιοχές. Θα πρέπει να δούμε και το κόστος ε, του δικτύου. Πάντως το μηχανολογικό κόστος του δικτύου είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τις ε, διαφορές ε, σε ό,τι αφορά την παραγωγικότητα και το δυναμικό ενέργεια των διαφόρων περιοχών. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική διάσταση που είπατε και το θέμα του λογαριασμού του ηλεκτρικού για τα νοικοκυριά. Έχουμε και εσωτερικές και εξωτερικές πτυχές. Και αν προσθέσουμε κάτι τώρα στο λογαριασμό που δεν υπήρχε πριν λόγω της μόλυσης, δύσκολο θα είναι να φανταστούμε ότι θα μειώνεται ο λογαριασμός. Να, μειωθεί ο λογαριασμός του, ηλεκτρισμού μάλλον αποκλείεται. Βέβαια δεν έχω καμιά κρυστάλλινη σφαίρα να μαντέψω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, αλλά μάλλον θα υπάρχει μια αυξητική τάση. Δεν μιλώ για το συνολικό οικονομικό κόστος, μιλώ για το τι θα πληρώνει ο καταναλωτής μάλλον θα πληρώνει περισσότερο. Κάτι που μας οδηγεί να αναζητήσουμε τις πιο φθηνές λύσεις για να εφαρμόσουμε τους ε, στόχους των πολιτικών μας. Γιατί αλλιώς ε, θα διονκώνεται όλο και περισσότερο αυτός ο λογαριασμός του ηλεκτρισμού και θα γίνει υπέρογκος και αδύνατο να πληρωθεί κάποια στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε μείωση κόστους χρειαζόμαστε, να βρούμε πιο ευρηματικούς, πιο έξυπνους μηχανισμούς. Αλλιώς δεν πρόκειται να ελοπίσουμε τους στόχους μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους δύο καλεσμένους μας και για την παρουσία τους και φυσικά για τις ε, παρουσιάσεις που μας έκαναν. Και να περάσουμε στο τελευταίο πάνελ, το τρίτο και τελευταίο πάνελ της ακρόασης αυτής. καλωσορίζοντας τους δύο τελευταίους καλεσμένους μας, δίνοντας τους αμέσως το λόγο, τον κύριο Όγκορσφερ από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Παρακαλώ πρώτα, εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, θα είμαι πολύ σύντομη και θα προσπαθήσω να ενσωματώσω ήδη κάποια από τα σχόλια, τις ερωτήσεις που ακούστηκαν νωρίτερα από πλευρά των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ξεκινώντας λοιπόν, θα θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται να σα παρουσιάσω και πάλι τον ενεργειακό δικό χάρτη. Είναι γνωστό, συνδεδομένο. ο στόχος είναι μείωση από 80-95% των εκπομπών δεξιού του άνθρακα για το 2020 είναι κάτι που έχουν αποφασίσει αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Στόχος κοινό σε όλη μας τη δουλειά, σε όλο το έργο που άλλωστε πρακτικά βλέπετε και σήμερα και, συγκρι... και από τόσο υπόθηκαν σήμερα, αλλά και συγκρινώντας με τόσο έχουν κάνει λοιποί παράγοντες, αλλά και στον ε, επιμέρου ε, χώρο, στα επιμέρου δηλαδή τη Γερμανία, Δανία κτλ. Εάν συνδυάσετε όλε τι προτάσει των εθνικών, τι εθνικέ προτάσει των κρατών μελών, δεν αποτελεί το άθροισμα του ε, ισοδύναμο του οδικού χάρτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Δηλαδή θα έχουμε τι εισαγωγέ από τι εξαγωγές. Και άρα χρειάζεται μια πιο σαφή εικόνα για την ενέργεια για το μέλλον. Χωρί να αποτελεί αυτό πρόβλεψη, μπορούμε, ασφαλή πρόβλεψη, μπορούμε να έχουμε, πρόγνωση καλύτερα, ε, μπορούμε να έχουμε μια σχετικά ασφαλή πορεία σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις και θέλω να δώσω και κάποια στοιχεία για το τι θα κάνουμε στα επόμενα βήματα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο ενεργειακός οδικός χάρτης σχεδιάστηκε με στόχους την ασφάλεια της προμήθειας, την ε, βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, αυτό το τρίγωνο των ε, στόχων, για το οποίο θα σας και παραδείγματα, αλλά όντως είναι πολύ σημαντικό και οι τρεις πτυχές να καλύπτονται στην πορεία για, το, για τη μείωση 95% Παράλληλα δηλαδή εξετάζουμε και τις αγωγές και τις εξαγωγές και τις τιμές και το κόστος των διαφόρων σενάριων που αναπτύσσονται. Ήδη παρουσιάστηκε ότι υπάρχουν διαφορετικά σενάρια για αποδέσμευση από τον άνθρακα. Το πρώτο σας στόχο έχει να καλύψει καταρχάς την κατάσταση όπως υπάρχει στα κράτη-μέλη. Πρώτος στόχος ήταν αυτός, με χώρες, παραδείγματι, που έχουν μεγάλη εξάρτηση ε, από τις με μεγάλη παρουσία των ανανεώσιμων, άλλε όπου έχει καθυστερήσει πολύ σύλληψη και ε, αποθηκευσή άνθρακα για διάφορους λόγους, ε, χώρες όπου δεν έχουν πυρηνική ενέργεια, γιατί σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει η καλή αποδοχή, αλλά όχι σε όλα, διαφοροποιημένη τεχνολογία προμηθειών και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα καταγράφουμε όλα για να δείξουμε πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το κόστος αλλά και το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών και βάσει βεβαίω των γνώσεων που έχουμε αυτή τη στιγμή στη θέση μα με την τεχνολογία ε, και με τα μοντέλα που έχουμε. Δηλαδή, ε, ασβεστολιθικό φυσικό αέριο δεν έχουμε περιλάβει, ούτε το αντίστοιχο πετρέλαιο. Ε, είναι κάτι που μας απασχολεί στις μελέτες μας και θα ενταχθεί ασφαλώς σε μελλοντικέ μελέτες, αλλά πέρσι που έγινε αυτή η έρευνα, η μελέτη μάλλον δεν ήταν πολύ πρόημο το να ενταχθούει και το ασβεστολιθικό φυσικό αέριο. Έχουμε όμως αποκεντρωμένες και κεντρικά οργανωμένες ανανόσιμες πηγές ενέργειας και άλλες λύσεις λάβει υπόψη. Για την ασφάλεια λοιπόν των προμηθειών. Σε κάθε σενάριο αποδέσμευση από τον άνθρακα μειώνεται η εξάρτηση από τις αγωγές, μειώνονται δηλαδή οι ενεργειακές αγωγές, απλώς και μόνο με την αποδέσμευση από τον άνθρακα, γιατί έχουμε λιγότερες αγωγές βεβαίως ορυκτών καυσίμων, ταυτόχρονα όμως και περισσότερες ανανεώσιμε πηγές, οι οποίες προέρχονται τουλάχιστον όσον αφορά το σενάριο το οποίο, στο οποίο εμείς έχουμε δουλέψει από το εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι τιμές στην ενέργεια που συζητήθηκαν και από το προηγούμενο πάνελ, είτε πρόκειται για αποδέσμευση άνθρακα είτε μη, ε, η πορεία είναι να αυξηθούν, ανάλογα και με την πολιτική του κάθε κράτους, αλλά πάντως και γενικά, μέχρι το 2030. Και βέβαια χρειάζεται να εξυγχρονιστεί να εξυγχρονιστούν υποδομές, να έχουμε φιότερα δίκτυα, να έχουμε καλύτερες υπερσυνοριακές διασυνδέσεις, ε, να εισεχάγουμε βέβαια τις ανανεώσιμες, αλλά και να εξυγχρονίσουμε, γιατί σε πολλά κράτη-μέλη είναι πεπαλαιωμένος ο εξοπλισμός και οι υποδομές και αυτό θα πρέπει να γίνει, όπως είπα, είτε με είτε χωρίς την αποδέσμευση από τον άνθρακα ε, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και βεβαίω πτήσετε το θέμα μετά ε, που θα πρέπει να λύσουν τα κράτη-μέλη του πώς θα χειριστούν τις μας. Επίσης από τη δουλειά μας καταλήγουμε στο συμπέρασμα Ε, να κοιτάξουμε το κόστος της αποδέσμευσης από τον άνθρακα. Δεν είναι πιο δαπανηρή βέβαια από την ε, ε, πολιτική που έχουμε τώρα, γιατί θα έχουμε λιγότερε εισαγωγέ το καυσιμών, όπως είπα. Όμως από την άλλη θα έχουμε κεφαλουχικές δαπάνες σημαντικές στην αρχή τουλάχιστον μέχρι την, εισαγωγή, την πλήρη εισαγωγή των ανανεώσιμων. Εν τέλει, το επόμενο βήμα. Ο ενεργειακός οδικός χάρτης θα πρέπει να συστηθεί και να ανοίξει το δρόμο για πιθανές επιλογές για την ενέργεια μακροπρόθεσμα. Αυτό πράττουμε δηλαδή σήμερα εδώ με την ακρόαση, αλλά και με άλλους φορείς εμπλεκόμενους και μέσα στα κράτη-μέλη. Προτεραιότητα είναι η παρακολούθηση και η υλοποίηση των στόχων του 2020, η μείωση των αέριων ε, θερμοκηπίου δηλαδή, οι ανανεώσιμες και η καλύτερη ε, αποτελεσματικότητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας. Η υλοποίηση της οδηγίας για την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας βεβαίως βοηθά και εκείνη στην εξοικονόμηση κατά 20% της ενέργειας. Αλλά όπως είπα, οι επενδύσεις είναι μακροπρόθεσμες και έτσι για το 2013 θα είμαστε ε, θα έχουμε στη θέσή μας μια μελέτη, μια προβολή για την περίοδο μετά το 2030 Γι' αυτό μα ενδιαφέρουν ιδιαίτερω οι αντιδράσει που βλέπουμε τώρα και για το ε, φύλλο πορεία στον οδικό χάρτη και για την αποδάσμευση από τον άνθρακα. Και βεβαίω τώρα λόγο θα κάνουμε και την ανάλυση μα ω προ του τρει στόχου μα. Και θα ε, επανέλθουμε με ένα ε, επικαιροποιημένο σενάριο που θα λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία για τις ανανεώσιμες του 2012, γιατί είχαμε ως έτο αναφορά στο 2009 μέχρι τώρα. Θα έχουμε λοιπόν και τις επαφές μας με όλα τα κράτη-μέλη και έτσι μέχρι τα το τέλη του τρέχοντος ή ίσως αρχές του προσεχούς έτους θα έχουμε ένα νέο σενάριο και την προετοιμασία για το πλαίσιο για μετά το 2030. Σαφές είναι, και κλείνω, αυτό το οποίο λέμε χωρίς πισωγυρίσματα, ανεξαρτήτως του σενάριου, ανεξαρτήτως των πολιτικών επιλογών και ξέρω ότι θα είναι διαφορετικές τα τη μερη χρειαζόμαστε πιο ευφύς υποδομές, χρειαζόμαστε ένα σημαντικό ποσοστό ανανεώσιμων πηγών και χρειαζόμαστε πολύ καλύτερη αποτελεσματικότητα στη χρήση ενέργειας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Γιανκόφσκι από το Witam Państwa bardzo serdecznie. Καλησπέρα σας. Βασικός στόχος της μου είναι να σας παρουσιάσω ε, τα αποτελέσματα που θα έχει ο ενεργειακό οδικός χάρτη του 2050 για την Πολωνία και για άλλες χώρες που απάδουν από τη γενική εκτίμηση. Ε, ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη για κάποιες αδυναμίες του εγγράφου. Ε, και θα προσπαθήσω να μιλήσω όσο πιο σύντομα γίνεται λόγω της κρίσης και του χρόνου. Ξεκινάμε λοιπόν από υπενθυμίζοντας τις μέχρι τώρα δράσεις. Ο στόχος ε, η μείωση εκπομπών τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. Έχουμε τη μείωση του 20% το βασικό στόχο, ενώ οι νέες προτάσεις μιλούν για το 80% μείωση μέχρι το 2050 κάτι που δημιουργεί τεράστιε προκλήσει για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μέχρι τώρα προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ε, προέβησαν σε κάποιε αξιολογήσει ε, των επιπτώσεων. Δυστυχώ είχαμε τις συνολικές εκτιμήσεις επιπτώσεων για το σύνολο της Ένωσης αλλά και για επιμέρους κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν όμως ολοκληρωμένες ε, μελέτες για τα επιμέρους αποτελέσματα στις διάφορες χώρες. Αυτό είναι ένα, ένα μείον της συζήτησης. Θα πρέπει να, να συμπληρώσουμε λοιπόν τη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αποτελέσματα μελέτες επιπτώσεων για συγκεκριμένες χώρες. Για παράδειγμα έχουμε την περίπτωση της Πολωνίας για την μελέτη αυτή χρησιμοποίησαμε ε, πρότυπα ε, που είναι πολύ αποδεκτά και από την πολωνική κυβέρνηση και κυρίως χρησιμοποίησαμε τρία σενάρια ε, με βάση το στόχο της μείωσης των εκπομπών. Έχουμε το φιλελεύθερο σενάριο, χωρίς δηλαδή περιορισμούς των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε το σενάριο της συνέχισης με την εισαγωγή του πακέτου των εκπομπών και το τρίτο σενάριο της ε, απαλλαγής από, τον άνθρακα με βάση τους στόχους για το 2050. Το βασικότερο, οι, βασικότεροι, οι βασικότερες υποθέσεις που χρησιμοποίησαμε ήταν αυτές που χρησιμοποίησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είχαμε τα αποτελέσματα για τέσσερις βασικούς τομείς. Για το σύνολο της οικονομίας, για τα νοικοκυριά, για τη βιομηχανία και για ολόκληρο το ενεργειακό σύστημα. Τα βασικά αποτελέσματα της πολωνικής μελέτης καλύπτουν μια, ένα ευρύ φάσμα δεδομένων. Για παράδειγμα, οι εκπομπέ διοξείδιο του άνθρακα μειώνονται και στα τρία σενάρια και κυρίω με το σενάριο τη απαλλαγή από το άνθρακα που έχουμε μείωση τη τάξη του 70% σε σχέση με, με το 1990. Βασικό αποτέλεσμα της κλιματικής πολιτικής στην Πολωνία είναι η αύξηση των ενεργειακών τιμών η απαλλαγή από την ενέργεια οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των τιμών σε σχέση με το πρώτο, το φιλελεύθερο σενάριο, χωρίς περιορισμό δηλαδή σε εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, ε, η, η πολιτική αυτή ε, επηρέασε και το θέμα της συμπαραγωγής ε, ηλεκτρισμού και, θε, και, και θερμότητας τα αποτελέσματα στην Πολωνία θα είναι πολύ πιο σοβαρά από το μέσο όρο τη Ένωση. Με το κλιματικό πακέτο και την αύξηση των ενεργειακών τιμών θα επιβραδυνθεί ο, οικονομικός, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης από το 2020 μέχρι το 2030. Μόνο μετά το 2030 διαπιστώνουμε κάποιες θετικές επιδράσεις εξαιτία της ε, μικρότερης εξάρτησης από τα ρηκτά καύσιμα. Έτσι θα έχουμε όμως ε, αύξηση των ενεργειακών πηγών και επιβράδυση της οικονομικής ανάπτυξης ε, πάλι μετά το 2040. Ένας πολύ σημαντικός ε, δείκτης είναι η συμμετοχή του κόστους της ενέργειας ε, στον προϋπολογισμό των οικοκυριών. Και στην Πολωνία σήμερα, στα μισά νοικοκυριά, το μερίδιο της, της, των ενεργειακών λογαριασμών είναι πάνω από 20%, πολύ ψηλότερο δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, το επίπεδο το 10% θεωρείται ως κατώτερο κατόφλι για την ενεργειακή ένδυα. Οι δείκτες λοιπόν μας δείχνουν ότι μόνο με το πρώτο, το φιλελεύθερο σενάριο μπορούμε να μειώσουμε το μερίδιο αυτό της ενέργειας στο λογαριασμό των οικοκυριών. Ενώ το τρίτο σενάριο της απαλλαγής από τον άνθρακα έχουμε, οδηγούμαστε σε αύξηση 14-15% ήδη από το 2020, κάτι που θα οδηγήσει σε ενεργειακή ένδυα τα πολωνικά νοικοκυριά. Η κλιματική πολιτική θα αυξήσει το κόστος και τη βιομηχανία. Κάτι που αφορά κυρίως το ε, έμεσο κόστος σε ό,τι αφορά την αγορά των αδειών για το σύστημα εμπορίας εκπομπών αλλά και το άμεσο κόστος ε, της αγοράς ενέργειας και τις, ε, τους φόρους για τον άνθρακα. Αυτά, αυτό το κόστος θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Και κυρίως η χημική βιομηχανία, η βιομηχανία, η χαλιβουργία, τα ορυχεία, τα δηληστήρια και η παραγωγή χάρτου θα επιβαρυνθούν περισσότερο από τις αυξήσεις των τιμών. Αυτές ε, οι βιομηχανίες επίσης απειλούνται κυρίως από το carbon leakage, από τη διαρροή του άνθρακα. Φαίνεται ότι απειλείται λοιπόν το 1 τρίτο της ε, ε, πολωνικής βιομηχανίας που απασχολεί 800.000 εργαζόμενους. Κάτι που θα, θα φέρει την Πολωνία σε δύσκολη ανταγωνιστική θέση απέναντι στην Ουκρανία και την Λευκορωσία που δεν δεσμεύονται από αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης, η επιρροή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην ενεργειακή πολιτική θα είναι τεράστια θα είναι διπλάσια από το κόστος κατασκευής εγκαταστάσεων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης θα αυξηθεί και το κόστος δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων γιατί χρειαζόμαστε τεχνολογίες που είναι πολύ πιο ακριβές. Επίσης θα αυξηθεί και το ετήσιο κόστος αν ε, θέλουμε να αυξήσουμε το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να οδηγηθούμε στο 20% της μείωσης, ενώ το κίτρινο είναι το κόστος μετά, μετά την εφαρμογή του στόχου του 80% της μείωσης. Βλέπετε το κόστος αυξάνεται με τα χρόνια, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερη καθυστέρηση στην εφαρμογή όλων αυτών των υποχρεώσεων. Παρά τη μείωση λοιπόν των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, θα αυξηθεί και το κόστος αγοράς των ε, αδειών ε, εμπορίας εκπομπών, αλλά και το κόστος ε, του φόρου άνθρακα. Ε, όλο, αυτό το, όλο αυτό το κόστος που θα είναι γύρω στα 9 δισεκατομμύρια το χρόνο θα έχουν αρνητικές επιρροές στη βιομηχανία. Έχουμε τα αποτελέσματα για την Πολωνία. Βέβαια έχουμε διαφοροποίηση ε, των δομών των ε, ορυκτών καυσίμων και της τεχνολογίας. Βέβαια τα πιο ε, σημαντικά αποτελέσματα είναι τα αρνητικά, πολύ πιο αρνητικά στην Πολωνία από ότι στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Θα διαρωτηθεί κανείς μήπως είναι υπερβολικά τα αποτελέσματα, μήπως είναι διωγγωμένα. Θα πρέπει όμως να δούμε και τις μελέτες Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνουν τα αποτελέσματα ανά κάθε χώρα. Βλέπουμε ότι στην Πολωνία η επιβαρύνση είναι πολύ μεγαλύτερη από τις υπόλοιπε χώρες από την ενεργειακή πολιτική που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το κλιματικό πακέτο, έχουμε ε, για για την απασχόληση, το ΑΕΚ και την κατανάλωση πολύ πιο αρνητικά αποτελέσματα από ότι ε, ο κοινοτικό μέσος όρος. Αυτές ε, οι τιμές προέρχονται μόνο από ένα τμήμα της εφαρμογής της κλιματικής πολιτικής. Επίσης, μια ανισότητα μεταξύ των κρατών δημιουργεί ο, οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί. Δημιουργούν οι, οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί από το πακέτο αυτό. Τρεις μηχανισμοί θα μειώσουν το κόστος εφαρμογής ε, του περιβαλλοντικού πακέτου στην Πολωνία. Βέβαια αυτό θα πρέπει ε, να γίνει μετά από τη λήψη απόφασης για την υλοποίηση αυτού του πακέτου. Βέβαια οι μηχανισμοί αυτοί απέτυχαν στην περίπτωση της Πολωνίας, κάτι που έδειξε η πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η μελέτη αυτή και οι δείκτες δείχνουν ότι είτε με μηχανισμούς αναδημετικούς είτε χωρίς αυτούς, το κόστος ε, εισαγωγής του ενεργειακού πακέτου και του περιβαλλοντικού στην Πολωνία θα είναι ε, πολύ μεγαλύτερο. Θα είναι διπλάσιο το κόστος για την Πολωνία από ό,τι για τον κοινοτικό μέσο όρο. Και ερχόμενο στα αποτελέσματα θα ήθελα να τονίσω ότι η κλιματική πολιτική δημιουργεί τεράστια απειλή και για το βιωτικό επίπεδο των Πολωνών, αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη της Πολωνίας. Η οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι η βασική υποχρέωση τη Πολωνίας απέναντι στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να κρατήσει τον ρυθμό οικονομική τη ανάπτυξη. Γι' αυτό και δεν αντιλαμβανόμαστε τι πιέσει που ασκούνται προ την Πολωνία να αισθενιστεί τέτοιου στόχου που θα δημιουργήσουν τόσο σοβαρέ απειλέ για την οικονομική τη ανάπτυξη. Και άσχετα με τι προηγούμενε παρατηρήσει, ο ενεργειακό ε, οδικός χάρτη, ούτω ή άλλω περιέχει κάποιε σοβαρέ αδυναμίε και η βασική αδυναμία είναι ο τρόπο ε, υπολογισμού των αποτελεσμάτων τη απαλλαγή από τον άνθρακα σε σχέση με το γενικό σενάριο για, τον περιορισμό των κλιματικών αλλαγών. Τι γίνεται σε περίπτωση που δεν, υλοποιεί, δεν ε, συναυθεί παγκόσμια συμφωνία για την μείωση των κλιματικών αλλαγών. Τι θα κάνει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα επίσης Ολοκληρώνοντας, να σας παραπέμψω στην λεπτομεριακή παρουσίαση που σας έχω μοιράσει. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Πρέπει να δώσω το λόγο και στην κυρία Τζαβέλα βεβαίως, άρα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Τζόρνταν, λιγότερο από ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. αναφέρατε ότι οι συζητήσεις αυτές θα αποτελέσουν, ε, θα ακριθούν και από το πολιτικό πλαίσιο. Αλλά είπατε ότι αναμένεται και νέους υπολογισμούς βάσει άλλων σενάριων. Μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτι περισσότερο. Τι εννοείται άλλα σενάρια, ποια είναι τα άλλα σενάρια και πότε μπορούμε να περιμένουμε τα νέα αυτά σενάρια. Υπάρχει, χρόνο, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Επίσης ε, είπατε ότι λάβατε υπόψη σας ε, το τρίγωνο της ε, αηφορίας. Κατά την άποψή μου όμως έχετε υπογραμμίσει κυρίως το, την περιβαλλοντική συνιστόσα. Δεν Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά την ανταγωνιστικότητα και δεν θυμάμαι πουθενά να αναφέρεται την απαλλαγή από τον άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στον υπολογισμό του ΑΕΠ δεν λαμβάνεται υπόψη το κόστος κλιματικής αλλαγής, ας πούμε τις μεγάλες αυξήσεις των πλημμυρών. Επίσης, στον υπολογισμό της, των αναγκών δεν λαμβάνεται υπόψη και το πρόγραμμα για την ενεργειακή αποδοτικότητα 2020, van Μπρέντ. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση για την την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπω να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στον δικό χάρτη και τα σενάρια που σε αυτόν περιέχονται και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πολωνικής ε, έκθεσης. Το κείμενο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βλέπουμε ε, βάσει του σενάριου ότι η απαλλαγή από εκπομπές άνθρακας δεν κοστίζει περισσότερο από την μία απαλλαγή. και βεβαίως εδώ θα ευγραμμιστώ και με την ερώτηση της ε, κυρίας Φιώνα, ε, γιατί βεβαίως ε, εάν δεν έχετε αναφέρει καθόλου το θέμα της μόλυνσης, ίσως αν μπει και αυτή η συνιστόσα τότε να εξισορροπηθεί καλύτερα η κατάσταση. Ναι. Ευχαριστώ κυρία Χίμπνερ. Όλοι αναφερθήκατε στην αύξηση της ζήτησης ενέργειας, άσχετα με τις πηγές. Έχουμε και την ε, χαμηλή αξιοπιστία των ε, ανανεώσιμων ποιών ενέργειας. Έχουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται και από τη δέσμευση αποθήκευση άνθρακα. Έχουμε μεγάλες απώλειες, έχουμε τα συμβατικά μέσα παραγωγής ενέργειας. Έχω όμως μία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγξε τον ε, την επιρροή που θα έχει αύξηση τη τιμή ενέργεια στην καθημερινότητά μα, γιατί θα είναι υψηλή οι λογαριασμοί ενέργεια. Πώ θα του καταβάλουν τα νοικοκυριά. Δεν πιστεύω ότι δεν θα αυξηθεί η ζήτηση. Πιστεύω ότι θα αυξηθεί η ζήτηση του ηλεκτρισμού. Εμείς μόνο για οικονομίες μιλούμε, μόνο αυτό μας ενδιαφέρει μέχρι το 2020-30. Αλλά τι γίνεται με την αποτελεσματικότητα των νέων καινοτόμων πολιτικών. Μόνο ε, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη και την αποδοτικότητα, ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ε, ζήτηση του ηλεκτρισμού και όχι απλώς να λέμε ότι δεν θα υπάρξει τέτοια αύξηση της ζήτησης. ήθελα να ευχαριστώ και τους δημιουργητές και να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν αλλάζουν σενάρια μέσα με τις άλλες δυνικές διευθύνσεις. Γιατί όλο και προς αν επικοινωνούν μάλλον τα σενάρια τους στις άλλες διευθύνσεις γιατί βλέπω όλο και περισσότερες αποκλήσεις μεταξύ των δικών σας προτάσεων και αυτών των άλλων γενικών διευθύνσεων. Και αντίστοιχα οι Υπουργοί των Οικονομικών δεν, είμαι, δεν φαίνονται να είναι διατεθειμένοι να ε, χρηματοδοτήσουν αυτές τις εξελίξεις. Έχετε λοιπόν κάποια επαλήθευση των προτάσεών σας από τις Γενικές Ευθύνσεις για τα Οικονομικά. Για τον Πολωνό κύριο. Έχετε κοιτάξει καθόλου ο καταναλωτή πώς το βλέπει το θέμα, ο Πολωνός καταναλωτή ο πολίτης. Τον ενδιαφέρει, ενδιαφέρεται πολύ, λίγο, καθόλου. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δύο λόγια μόνο. Η Επιτροπή εργάζεται συλλογικά. Όλοι οι οδικοί χάρτες 2050 κυρίως Γενική Διεύθυνση Κλίματος, Μεταφορών Ενέργειας, αλλά και η ΛΥΠΗ ε, για το ΑΕΠ, για τον πληθυσμό, μακροοικονομικό σχεδιασμό, επιχειρήσεις, ε, βιομηχανία, ε, όλες οι σχετικές αρμόδιες υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνεργάζονται και είναι κάτι το οποίο κάνουμε μάλιστα τακτικά, δηλαδή κάθε δύο-τρία χρόνια πρέπει να επικαιροποιούνται τα στοιχεία της πολιτικής, η βάση δηλαδή της πολιτικής και η εξέλιξη των τιμών και αυτό βέβαια σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τα υπουργεία τους. Άρα υπάρχει. Ασφαλώς υπάρχουν τι συζητήσει, αλλά εν τέλει καταλήγουμε σε μια κοινή θέση γιατί πρόκειται για μια κοινή επιχείρηση ως προς τις διαφορές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχουν πτυχές της αξιολόγησης ε, επιπτώσεων που δεν ελήφθησαν υπόψη σε αυτή τη ε, μελέτη της Πολωνίας. Καλύπτουν κάποιες πτυχές αλλά όχι το κόστος από την κλιματική αλλαγή και Φαντάζομαι θα αντιδράσει ο κύριο από την Πολωνία, αλλά πάντω πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχουν θετικέ, θα υπάρξει θετικό αντίκτυπο και στι θέσει εργασία. Δηλαδή, μπορεί από ένα τομέα να χαθούν θέσει εργασία, αλλά μπορεί να κερδιθούν πολλέ σε άλλον, όπω πράσινε θέσει εργασία, τοπικέ τεχνολογίε, νέε τεχνολογίε κ.ο.κ. Αυτό το δείχνει και η δουλειά τη Επιτροπή. Και επίση Πρέπει να επισημάνω ότι και εμείς έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή ανάλυση κατά τη ε, μελέτη των προγνώσεων για την αποδέσμευση από τον άνθρακα, λαμβανόμενη υπόψη την ιδιαιτερότητα των κάθε κράτους μέλους. Και ναι, θέλουμε να εστιαστούμε ως προς τη διαχείριση της ζήτησης, ως προς την αποτελεσματικότητα της ενέργειας, ως προς την ενημέρωση του καταναλωτή, ω προ τη δυνατότητα για αλλαγή, παρό, για αλλαγή παρόχου, για το κόστο και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που συμφωνώ βεβαίω είναι ε, πάρα πολύ σημαντική για τον καταναλωτή. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ, ο κύριο Ιακώβσκι. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση. Οικονομίες και ενεργειακή αποδοτικότητα. Εμείς ε, στο σενάριό μας είδαμε ότι έχουμε πενταπλάσια αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Και ε, είναι τεράστια ε, η αύξηση της ε, ενεργειακής αποδοτικότητας. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν το λάβαμε αυτό υπό, υπόψη. Είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή η ενεργειακή αποδοτικότητα που χάνουμε από τον κοινοτικό μέσο όρο σε ό,τι αφορά τις ε, διαφορέ μεταξύ της εκτίμησης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της πολωνικής μελέτης. Απ' τη μια υπάρχουν ε, κάποιες αποκλησει αλλά υπάρχουν και κάποιες συγκλησει ε, και κοινά σημεία. Για παράδειγμα, το προτινόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σενάριο δείχνει μία, ένα, ένα συστημικό αύξ, μια ενα συστημικο συστημικη αυξηση των, του ενεργειακού κόσμου από 10 προς 14%. Κάτι που δείχνει ε, η, τη δυσκολία πρόσβασης ε, ε, των των οικοκυριών στην ενέργεια. Και επειδή το μέσο εισόδημα στην Πολωνία είναι πολύ χαμηλότερο από το κοινοτικό μέσο όρο, μια τέτοια αύξηση των ενεργειακών τιμών θα είναι πολύ πιο επώδυνη για τα πολωνικά νοικοκυριά. Τώρα για τις υπόλοιπες διαφορές, σε μερικές περιπτώσεις είναι δύσκολη η σύγκριση. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το συστημικό κόστος δίνονται οι μέση όροι για το 2050, αλλά δεν ε, υπάρχουν συγκεκριμένες αξιολογήσεις ε, για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Στον οδικό χάρτη για το 2050 δεν δίνονται τα συστημικά κόστη της ενέργειας, οπότε είναι πολύ δύσκολο να συγκρίνουμε τις τάξεις μεγέθους των διαφόρων σενάριων, λαμβάνοντας υπόψη ότι το σενάριο fragmented action της κατακαιρματισμένης δράσης λαμβάνεται υπόψη μόνο στο roadmap ε, του 2050, ενώ στον ενεργειακό χάρτη, ε, ε, οδικό χάρτη δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στη, με, στη μελέτη της το μέσο όρο. Εμείς ασχολούμαστε με την πολωνική κατάσταση, οπότε και εδώ οι τάξεις μεγέθους δεν είναι εύκολα συγκρίσιμες. Υπάρχουν λοιπόν, επαναλαμβάνω, και ομοιότητες και διαφορές. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση στην Πολωνία είναι πολύ διαφορετική από τον κοινοτικό όρο, γι' αυτό και τα αποτελέσματα της πολωνικής μελέτης είναι πολύ διαφορετικά από τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ τους συζητητέ. Η κυρία Τζαβέλα για να ολοκληρώσουν να ολοκληρώσει τις εργασίε μας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους ε, συμμετέχοντες ε, και τους ε, ομιλητές που έκαναν τις παρουσιάσεις τους και τους συναδέλφους που παρακολούθησαν. Θα θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Αυτή η έκθεση πρέπει να αναφερθεί στην ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να το υπενθυμίσω αυτό στους συναδέλφους στην Επιτροπή Ήτρε. Κοιτάξτε, εδώ δεν ασχολούμαστε με την κλιματική αλληγή. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε, να καταρτήσουμε την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι πολύ ασαφής, ενώ οι πολίτες, η βιομηχανία, οι επενδυτές ε, είναι ιδιαίτερα μπερδεμένοι σχετικά με το ποια είναι τελικά αυτή η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέω και το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω έτσι ώστε να το καταλάβουμε όλοι. Ε, η κλιματική αλλαγή είναι ένα ξεχωριστό θέμα. Εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε τώρα για την ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα ο δρόμος προς ε, την κατάληξη της ενεργειακής πολιτικής ε, θα είναι μακρύς. Ε, αναμφισβήτητα επίσης θα χρησιμοποιηθούν όλες οι μορφές ενέργειας ε, έτσι ώστε να επιτύχουμε τους ε, στόχους ε, που είναι ενεργειακή αποδοτικότητα, σωστή ανταγωνιστικότητα και τελικά επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και η γεωθερμία και η πυρηνική ενέργεια, αιωλική ενέργεια, η ενέργεια από τον ήλιο, αλλά και οι παραδοσιακές μορφές ενέργειας. Όλες μπορούν να παίξουν ρόλο, να μην το με αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή στην ακρόαση και ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Πρόεδρο για τον τρόπο με τον οποίο διεξήγαγε αυτήν την ακρόαση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Τζαβέλα, σας ευχαριστούμε όλους. Ε, ολοκληρώνουμε αυτό το τμήμα της συνεδρίασής μας, αλλά θα πάμε στο 2Q2, ε, εκεί δηλαδή που μέχρι τώρα συνεδρίαζε μόνη της Επιτροπή Μεταφορών, έτσι ώστε να ε, συζητήσουμε μαζί με τους συναδέλφους της Επιτροπής Μεταφορών θέματα που σχετίζονται και με την ενέργεια και που ενδιαφέρουν και εμάς. 2Q2 λοιπόν, ευχαριστώ.